Uh, Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, It's five past three. So. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Καταρχήν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην απογευματινή συνεδρίαση. Έχουμε και κάποιους επιπλέον συναδέλφους εδώ για την πρώτη συζήτηση της έκθεσης του κυρίου Τεραμπέλα, εκ μέρους της Επιτροπής για τις ε, οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων. Έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας για αυτή τη συζήτηση, γιατί προβλέψαμε μια μισή ώρα γιατί αισθανθήκαμε ότι θα ενδιαφέρει πολύ του συναδέλφου να συζητήσουν την πρόταση αυτή και στη συνέχεια από τις 4.30 ως ε, τις 5.30 ε, θα δούμε την έκθεση του κ. Κοφεράτη για τις συντάξεις ε, ως τις 5 με συγχωρείτε και στις 5 θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Καλωσορίζω και όσους μας ακούνε από το διαδίκτυο για τη συζήτηση για τις δημόσιες συμβάσεις. Ε, τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω να ε, θέλετε ένα αντίγραφο του newsletter. Μπορείτε να γραφείτε στην ιστοσελίδα μας και θα σας στείλουμε αυτό το newsletter όπου θα δείτε και όλη τη δουλειά της Επιτροπής μας και να ευχαριστήσω την προσοχή των συναδελφών των μελών της Επιτροπής μας ε, στο εξή. Ε, Σα έχω διανύμει το σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπή για την ε, Ενία πράξη της αγοράς. Ο κύριος Μπερνιέ, ο αρμόδιος Επιτρόπης για την Αγορά, μας ζήτησε να συνεισφέρουμε στο έργο του για το πρόγραμμα της Ενέας Πράξης για την Αγορά για το 2013. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο πρότασης και 89 τροπολογίες ε, θα ψηφίσουμε αύριο, θα περάσουμε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο και την Τετάρτη της Ολομέλειας και ο κύριος Μπερνιέ θα μας παρουσιάσει μια έκθεση για την εφαρμογή του Single Market Act. Μια πρόταση για το πώς θα βελτιωθεί η διακυβέρνηση της ε, ενιαίας αγοράς και τις ιδέες του για την πράξη για την ενιαία αγορά για το 2013. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ όσοι θα παρευρίσκεστε στο Στρασβούργο σημειώστε το με κεφαλαία στο ημερολογιό σα, στην ατζέντα σας ε, και θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους παρευρισκόμενου την Τετάρτη για να ακούσουμε τις προτάσεις του κυρίου Μπαρνιέ. Λοιπόν, όπω όλοι γνωρίζετε, μία από τι πιο σημαντικέ ε, προτάσει στο επί των οποίων εργαζόμαστε τώρα συνδέεται με τι ε, οδηγίε για τι δημόσιε συμβάσει. Ε, ο κύριο Ταραμπέλα είναι ο συγητής μα έχει εκπονήσει αυτή την έκθεση που είναι διαθέσιμη σε όλε τι γλώσσε. και έχουμε του κοιόδη που θα συνεισφέρουν. Νομίζω ότι ο κ. Βαντεκάπ θα μιλήσει εκ μέρου του κ. Έγγελ, ο κ. Κρόιτσμαν, τον ξανακαλωσορίζω σε αυτή την επιτροπή για τους φιλελευθέρους, ο κύριο Ρίλε για τους πρασίνους, ο κύριο Κόζουσνικ ε, για τη δική μου ομάδα και εγώ θα υποστηρίξω λίγο αργότερα, ο κύριος Ντεγιόγκ δεν είναι εδώ, ίσως να έρθει αργότερα. Έτσι λοιπόν, ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τραμπέλα σε λίγο, όμως να πω ότι αφού ακούσω τον κύριο Ταραμπέλα πρέπει ε, να συναντήσω τους Ιαπωνέζους γιατί συμμετέχω στην αντιπροσωπεία με την Ιαπωνία. Θα με αντικαταστήσουν λοιπόν στην Προεδρία. Έτσι λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Ταραμπέλα για να παρουσιάσει την έκθεσή του στην Επιτροπή. Merci. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μάλκολ. Καταρχήν αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι αυτή η έκθεση είναι ογκώδης και ε, όπως είπατε είναι μια πολύ εμβληματική έκθεση εξού και δεν χρειάζεται να δικαιολογηθώ σχετικά με την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και θα ήθελα μαζί σας να ε, εξετάσω διάφορες πτυχές από προτάσεις και να σχολιάσω τις προτάσεις της Δανικής Προεδρίας που μας ενέπνευσαν στο Κοινοβούλιο για ρήτρε που εστιάζονται σε ορισμένα θέματα. Δεν θα αναφερθώ σε όλες, αλλά βεβαίως θελήσαμε με μονομένα, ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, αυτό είναι ο ρόλος μας, να κάνουμε παραλληλισμούς και να δούμε πού είναι οι διαφορές με το Συμβούλιο άπαξ και αποφασίσουμε και προχωρήσουμε επί του θέματος. Κατόπιν ε, λοιπόν των διαδικασιών του πρώτου κλάστερ ε, και ε, εάν υπάρξουν νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φανούν σαν να επιβαρύνουν το θέμα στο μέλλον θα πρέπει ο επιλέγων να τον μειοδότη στον διαγωνισμό να μπορεί να ε, κινηθεί και γι' αυτό η απόδοση των συμβολέων πρέπει να μας απασχολήσει και μέσω του άρθρου 24 τονίζω την υποχρέωση για όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία ενώ διαφορετικά σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια των κρατών εάν θα προχωρήσουν ή όχι. Ένας από τους, βασικούς ε, στόχους της ε, ε, αναπτύξεως μέχρι το 2020 είναι αυτό και ε, εντείνει και την συνεργασία για την καινοτομία. Όσον αφορά το δεύτερο κλάστερ της δημόσιες αγορές, της δημόσιες προμήθειες σχετικά με τα άρθρα 64, 66, 67, 70 ουσιαστικά αναφερόμαστε στις τεχνικές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 40 για μια αηφόρο ανάπτυξη. Και αυτές οι νέες διατάξεις, οι οποίες είναι συνεκτικές, θα επηρεάσουν την δυνατότητα επιλογής του μειοδότη και θα έχουν διάφορες επιπτώσεις σχετικά με τις ε, υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται. Εντείνεται έτσι ο στρατηγικός ρόλος των αγορών όπως χρειάζεται και ε, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να, ε, του οποίου πρέπει να αμελήσουμε τη σημασία. Έχει τριπλή σημασία. Περισσότερη ε, προστασία για τους ε, εργαζομένους, μεγαλύτερη σαφήνεια, οικονομική και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Υπάρχει επιπλέον μεγαλύτερη διαφάνεια διότι πρέπει να υπάρξουν κριτήρια σαφή και υποχρεωτικά και στον ε, αναθέτοντα τον, ε, τον κριτή του διαγωνισμού ανατίθεται ένα πολύ ε, δύσκολο έργο και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα παραρτήματα 12, 13, 14 ιδίω που αναφέρονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν γνώση όλων των κοινοποιήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πράξης πλατφόρμας αντί τώρα να ψάχνουν δεξιά και αριστερά για κατακαιρματισμένες δημοσιεύσεις. Ε, όλες οι πληροφορίες λοιπόν οι ευαίσθητες ε, ε, πληροφορίες ούτως ή άλλως είναι σε ψηφιακή μορφή και ως εκ τούτου έτσι θα καταργηθούν ορισμένες ασφάλειες, ε, ε, ε, ασάφειες, ένα μεγάλο μέλος της γραφειοκρατίας και θα ξέρει κανείς ακριβώς εάν έχει τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει σε έναν μειοδοτικό διαγωνισμό δημοσίων προμηθειών ή όχι. Θα μειωθεί έτσι και το κόστος και το γραφειοκρατικό βάρος θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα ε, θεσπιστεί η αρχή best value for money, δηλαδή ε, να έχει καλή στην καλύτερη δυνατή απόδοση της επενδύσεώς του. Εξού και στα βασικά σημεία που τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προώθησα ε, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εξασφάλισαν μεγαλύτερη μεγαλύτερο ανταγωνισμό και ε, επέτρεψαν να ε, κατανεμηθεί καλύτερα η αγορά και στο άρθρο 16 που αναφορόμαστε στα κονσόρτσια για συγκεκριμένες χώρες και ιδίως στην Ιταλία βλέπουμε ότι ο θεσμός αυτός είναι αποτελεσματικός και χρήσιμος και στο άρθρο 44 η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει καλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διότι διευρύνεται το μέγεθος της αγοράς και επιτρέπει επιτρέπει στο μειοδότη να ε, καλύψει και να κερδίσει ε, την, ε, το διαγωνισμό και αυτό που είναι βασικό για μένα επίσης είναι η υπεργολαβία η οποία έχει θεσπιστεί σε πολλά κράτη-μέλη η Ιταλία είναι πολύ πιο αυστηρή από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γαλλία πληρώνεται κατευθείαν ο υπεργολάβος αλλά ο βασικός στόχος είναι να αποφύγουμε να διεισδύσουν οι εγκληματικές, τα διεγκληματικά δίκτυα σε αυτές τις διαδιακασίες και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζει κανείς τους, τους υπεργολάβους, να μπορεί να τους ελέγξει και μου έχουν λεχθεί πολλές περιπτώσεις για εργαζόμενους παρανόμους οι οποίοι αναλαμβάνουν τέτοια συμβόλαια χωρίς κανένα συμβόλαιο, καμία κοινωνική προστασία και αντιλαμβάνεστε ότι μέσω της προτάσεώς μου προσπαθώ βεβαίως να διατηρήσουμε την υπεργολαβία που είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα και όταν είναι υγιής πρέπει να διατηρηθεί γιατί επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε αγορά, αγορές που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να προσεγγίσουν αλλά δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική υπεργολαβία δηλαδή 7ο-8ο κλιμάκιο 7ο-8ο ε, υπεργολάβος κάποιος δηλαδή πήρε μία απλούστατα προμήθεια δεν εργάστηκε και δεν σεβάστηκε καμία νομοθεσία και νομίζω ότι εκεί χάνονται τα χρήματα και πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγιάνουμε όλο αυτό το δίκτυο και η υπεργολαβία να είναι αποτελεσματική και η είσοδος για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σε δημόσιες ε, αγορές και σε δημόσιες προμήθειες εκ των οποίων αποκλείονται από, μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με τα άρθρα 84, 85 και 87 χρειάζεται έλεγχος για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε σωστά την νομοθεσία στους διάφορους τομείς ε, δημοσίας υγείας, ε, κατανομής των δαπανών και αναλόγως των ε, κρατών. Είναι διαφορετική η κατάσταση, αλλά δεν θέλουμε να ενισχύσουμε τη γραφειοκρατία. Αντιθέτως, να υπάρχει πιο αποτελεσματικός έλεγχος. Όπου δεν υπάρχει λοιπόν ο οργανισμός ελέγχου των δημοσίων προμηθειών και των δημοσίων διαγωνισμών θα πρέπει να δημιουργηθεί. Και σε μεσογειακές χώρες όπως το Βέλγιο ή τη Γερμανία δεν χρειάζεται να ε, αναθεωρήσουμε το ισχύον καθεστώς όταν υπάρχει ήδη ένας ελεκτικός οργανισμός όποιος και να είναι είτε ε, υψηλότερου επίπεδου ή χαμηλότερου λόγω του ομοσπονδιακού χαρακτήρα θα μπορεί κανείς να συναλλαγεί με τις ισχύουσες αρχές. Θα ήθελα λοιπόν έως ε, προτού να να καταλήξω να σας πω στο σημείο 8 και 9 έχουμε την γενική οδηγία και στη συνέχεια τις τομέακες και έχω απλώς να σας πω ότι ό,τι ε, υπεραμείνομαι στη μία περίπτωση ε, θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στις δύο ε, και στη δεύτερη εκτός από το άρθρο 11β το όπου όπως τα ταχυδρομεία υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ε, η επιχείρηση δεν δημοσιοποιεί ε, την, ε, τον διαγωνισμό για να μην αποκαλύψει τη στρατηγική της συγκεκριμένα για τα ταχυδρομεία αλλά από εκεί στο να διευρύνουμε σε όλο το εύρος της οδηγίας δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτά τα άκρα και να εφαρμόσουμε την νομοθεσία και τα σχετικά άρθρα έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν δημόσιες οργανώσεις των οποίων η δραστηριότητα υπόκειται σε ανταγωνισμό και για στρατηγικές αγορές δεν θέλουν να αποκαλύψουν τις στρατηγικές τους εφόσον ο άμεσα ομόλογός τους του ιδιωτικού τομέα δεν το πράττει. Τέλος θα ήθελα να χαιρετήσω τους σκιώδη εισηγητές με τους οποίους συναντήθηκα επανειλημμένος. Ξέρω ότι σήμερα υπάρχει ένα Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητος και εκπροσωπείται μεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά θα πρέπει συγχρόνως να, διε... να κοπεί στα δύο και να παρακολουθεί και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητος. Όταν λοιπόν υπάρχουν ερωτήσεις προσπάθησα να απαντήσω στους συναδέλφους με την ιδέα των κλάστερς είτε όλους μαζί είτε ε, μεμονωμένα και ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ διότι με βοήθησε στην δύσκολη αυτή η εργασία με ένα πολύ στενό χρωμοδιάγραμμα και σας το λέω αυτό για όσους έχουν αναλάβει γνωμοθωτήσεις ορισμένοι λέγουν ε, ε, αυτοί μας ζητούν κάτι για χθες οι τροπολογίες λήγουν στις 14 Ιουνίου και μετά θα υπάρξουν οι γνωμοδοτήσεις. Υπήρξε όμως ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο προσπάθησα να σεβαστώ και αν αυτό ενοχλεί ορισμένους με στενοχωρεί αλλά προσπάθησα να συναντήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές και τους εισηγητές των γνωμοδοτήσεων και ευχαρίστως να υπάρξουν και άλλες διότι συζητάμε από τις 21 Δεκεμβρίου, τέσσερις σχεδόν πέντε μήνες με διάφορες συνεδριάσεις και δεν είμαστε στην αρχή, είμαστε όλοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν τονίσει τις διάφορες πτυχές και θα δούμε όταν θα κατατεθούν οι τροπολογίες τι γίνεται. Πρέπει όμως να σας πω ότι η μέθοδος μου εργασίας είναι να διαβουλεύομαι μαζί σας, να είμαι ανοιχτός σε όλες τις ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δεν αλλάζω πορεία. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και είμαι στη διάθεσή σας για τους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να κάνουν παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και για την διεξοδική αυτή πλήρη έκθεση. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εργασία σας και τη συνεργασία σας με τους σκιώδεις ηγητές. Όπως είπατε και εσείς, ακολουθούμε ένα χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί ουσιαστικά και τις οικονομικές απαιτήσει οι οποίες διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι περιμένουν να δουν την έκβαση αυτή τη έκθεση. Θα ακούσουμε τους κοιόδης ηγητές. Θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από τη Σουηδία. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ έχει καλέσει την ομάδα αυτή. Ελπίζω ότι χαίρονται τη συζήτηση για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα σήμερα το απόγευμα. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τους σκιώδεις συγητές Η κυρία Πετικάνινγκ Βάισερ, ε, ναι. Η κυρία Ρούλ επίση είναι στον κατάλογο, η κυρία Στάιλερ. Θα ακούσουμε καταρχάς πρώτα όλους τους πιο ηγητές, τον κύριο Κάμπα, Κρότσμαν, Ρούλερ, Κοζουσνίκ, Γιόγκα και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διαθεσή μας για να κάνουμε πλήρη συζήτηση. Οποιοδήποτε άλλος λοιπόν θέλει να πάρει το λόγο, ας μου το πει. Κύριε Βάιλερ. Με τον κύριο Βάντενκαπ θα ξεκινήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κατά των αρχών μου θα εκφραστώ στα αγγλικά σήμερα, γιατί ουσιαστικά αντικαθιστώ τον κύριο Φρανκ Έγγελ, σκιώδη ηγητή για το ΕΛΚΑ. Μην κατηγορείτε λοιπόν εμένα, αλλά κατηγορήστε αυτόν Βασικός στόχος αυτής της οδηγίας είναι η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των δημοσίων χρημάτων και γι' αυτό αποτελείται μια πολύ αποτελεσματική νομοθεσία όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 20% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να επιτευχθεί αυτό μέσω της απλούστευσης των κανόνων, όσον αφορά τον, τις διαδικασίες μειοδοτικών διαγωνισμών, τη βελτίωση της νομικής ασφάλειας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαδικασία αυτή και θα πρέπει βέβαια να προωθηθούν και κάποιες καινοτόμε λύσεις και να υπάρξει και μια βελτίωση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ακριβώς το εξήγησε και ο εισηγητής. Ο κύριος Σέγγελ είναι υπέρ του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Μάρκ Ταραμπέλα και σε πολλά σημεία συμφωνεί με τη γραμμή που ακολουθεί ο εισηγητής ιδίως την πρόθεση να υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για τη συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων για την ε, ανάθεση πάνω των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται. Η πρόταση της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολείται με την επέκταση και την ε, εμβάνθυνση των περιβαλλοντικών κριτηρίων, αλλά δεν θέτει πολλά κριτήρια όσον αφορά την κοινωνική διάσταση. Προκειμένου να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ο εισηγητής έχει χρησιμοποιήσει μια νέα έννοια κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία παραγωγής. Και μέσω της νέας αυτής έννοιας προβλέπει τη δυνατότητα συμπερίληψης κοινωνικών κριτηρίων στην ανάθεση και στην επιλογή. Ο κύριος Σέγγελ είναι σαφώς υπέρ της εξέτασης των κοινωνικών κριτηρίων στη διαδικασία ανάθεσης, αλλά δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη συμπερίληψη των κριτηρίων αυτών στα κριτήρια επιλογής. Γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μία επιλογή εταιριών οι οποίες ουσιαστικά θα, συν... θα κάλυπταν μόνο τα κριτήρια της περίφημης κοινωνικά βιώσιμης παραγωγής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα κριτήρια τελικά θα είχαν να κάνουν μόνο με την πολιτική που η εταιρεία αυτή και δεν θα υπήρχε άμεση σχέση με το υποεξέταση αντικείμενο κάθε φορά. Η κοινωνική αυτή διαδικασία παραγωγής που προτείνει ο εισηγητής θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά ως νέα έννοια. Είναι πολύ ασαφή η έννοια αυτή αυτή τη στιγμή όπως την προτείνει ο εισηγητή και θα οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα. Θα οδηγήσει για παράδειγμα στην εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων ως βασικό κριτήριο προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν ή να, να δοθεί, να παρασχεθεί μια υπηρεσία. Αυτές οι συλλογικές όμως συμφωνίες θα μπορούσαν ε, να εξεταστούν ε, μόνο αν είχαν ουσιαστικά δεσμευτική δύναμη σαν αυτή που έχει ένας νόμος και αν είχαν γίνει ουσιαστικά σφαιρικά αποδεκτές. Ο κύριος Σέγγελ δεν είναι κατά της διαδικασίας κοινωνικά βιώσιμης παραγωγής επί της αρχής, αλλά έχει κάποιες βάσιμες αφιβολίες ως προς τον ορισμό που χρησιμοποιείται και ως προς τη συμπερίληψή του σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάθεσης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει η έννοια αυτή να γίνει καταρχάς νομικά βιώσιμη και εφαρμόσιμη, προκειμένου να μην χαθεί η δυνατότητα σωστής και κατάλληλης ανάθεσης στα πλαίσια μιας δημόσιας σύμβασης. Στο άρθρο 71, ο εισηγητής προτείνει ένα σύστημα κοινή ευθύνης, προκειμένου να καλυφθεί όλη η αλυσίδα υπεργολαβίας. Ο κύριος Έγγελ είναι κατά ενός τόσο αυστηρού άκαμπτου συστήματος, γιατί ουσιαστικά θα επέδιδε ευθύνε στους βασικούς αναδόχους που δεν μπορούν στην πραγματικότητα να ελεγχθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης, το σύστημα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά σε πιο πολύπλοκα προϊόντα και πιο πολύπλοκες υπηρεσίες ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν εντελώς αφαίρετο και δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Συντοπεί ο κύριο Σέγγελ τι ανησυχίε του συγητή, ωστόσο πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες, κάποιοι βιώσιμοι περιορισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς όμως να βασιζόμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα φαντασίας. Η επέκταση της ε, χρήσης του πιο οικονομικού συμφέροντος ε, της πιο οικονομικής συμφέρονσης ανάθεσης είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει ο κύριος Έγγελ μολονότι θα πρέπει για τα υψηλά τυποποιημένα προϊόντα να μπορεί να χρησιμοποιείται και η αρχή της χαμηλότερης τιμής θα υποβάλει κάποιες τροπολογίες προκειμένου να υπάρχει ένα πιο ελαφρύ καθεστώς δημόσιας σύμβασης κάτω από το υφιστάμενο κατόφλι, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά. Όσον αφορά τώρα τις παραγράφους που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση, ο κύριος Έγκελ συμφωνεί με την προσέγγιση του εισηγητή, δηλαδή να τεθούν κάποιες αρμοδιότητες σε ορισμένα κράτη-μέλη και να αποφευθεί γενικότερα η υψηλότερη αύξηση του άχθους για συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Στο σχέδιο έκθεσης βέβαια έχουν καταβληθεί πολύ σημαντικές προσπάθειες από τον κύριο Ταραμπέλα. Οι προτάσεις αυτές ε, επαρκούν για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα γίνουν όμως και άλλες ανταλλαγές απόψεων προτού πούμε ότι έχουμε καταλήξει τελικά σε ένα τελικό κείμενο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για τα κομψά αγγλικά σας. Και τα εκτιμήσαμε ιδιαίτερα. Κυρίως ε, καθώς ε, εμείς πλησιάζουμε στο 60 επέτειο της ε, διαδοχή της Βασίλισσας στο θρόνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο Ταραμπέλα, ο οποίος προσπάθησε να να αλλάξει τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τέτοιων τρόπων ώστε να ενισχυθούν τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και άλλα θέματα που τον απασχολούν. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ε, ότι οι προσπάθειές του είναι εστιασμένες για να επιτύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και όπως είπε ο κύριος Ταλαμπρέλα, αν είμαστε φιλελεύθεροι ε, και έχουμε συγκεκριμένες ιδέες πρέπει να δούμε αν είναι λογικές οι προτάσεις και δεν θέλουμε γενικές απλώς δηλώσεις διότι σε μία ανάθεση μίας, ε, ενός έργου μετά από διαγωνισμό πρέπει να ξέρει κανείς εάν ε, ο εργολήπτης είναι σε θέση να εκτελέσει το έργο εάν πρόκειται να υπάρχει επικοδομητική εξέλιξη και γι' αυτό υπάρχουν διάφορα θέματα ε, τα οποία πρέπει να τονιστούν περισσότερο. Είπε ο κύριος Ταραμπέλα ότι πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά κοινωνικά κριτήρια σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, οπότε όμως θα υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και ανασφάλεια ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφερθεί ε, στο θέμα αυτό μόνο στην διανομή των φυλαδίων ενώ υπάρχουν ρυθμίσεις τα οποία ενιαία, ε, ενιαία πρόκειται να ρυθμιστούν όπως είναι η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργατείας. Πρέπει ε, επίσης να, να δούμε πώς θα λύσουμε και άλλα θέματα. Η, τρεις, η, διαφοροποίηση σε τρεις τομείς θεωρούμε ότι είναι υπερβολωθή και θα πρέπει να βοηθήσουμε τον εργολήπτη στα κρατη μερη για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απ' την άλλη πλευρά ο κύριος τα θέλει να ε, καταστεί υπόλογος ο καθένας που εμπλέκεται σε αυτή την αλυσίδα αλλά ε, αυτό θα πρέπει ε, επίσης να ισχύσει για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να στραφούν στους υπεργολάβους τους και τότε οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να κινηθούν τόσο εύκολα. Είναι, εύκολο, είναι σαφές ότι ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να σέβεται τα συμπεφωνημένα και ε, την νομοθεσία και αν αυτό δεν συμβεί πολύ σωστά είπε ότι ο κύριος ε, είπε ότι θα πρέπει να μπορεί να αποκλειστεί μία επιχείρηση αλλά θα πρέπει ε, να αποδειχθεί αυτό από έναν εξάρτητο δικαστήριο δεν φτάνει απλώς η κατηγορία και επίσης η ανάθεση των δημοσίων έργων είναι ευγενής στόχος αλλά επιπλέον θα πρέπει να γίνει με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο και άλλωστε ο κύριος Ταραμπέλα διαγράφει το θέμα των διατάξεων που αναφέρονται στις τις υπεργολαβίες ενώ θα πρέπει όπως ε, στην ε, οδηγία υπηρεσιών να συμμορφωθεί κανείς με την χώρα που είναι ο στόχος. Ε, δηλαδή θα πρέπει όλη η διαδικασία να είναι διάφανη και να δούμε βάσει ποιων αρχών γίνονται οι προκηρύξεις, διεξάγονται οι διαγωνισμοί και η επιλογή του ε, Επίσης ε, ε, ο κύριος Ταραμπέλα είναι αντίθετος σε ορισμένες αρχές της εσωτερικής αγοράς ε, που λέει ότι πρέπει να προστατεύσουμε το χώρο της παραγωγής και να μην υπάρχει προστατευσισμός ο οποίος μπορεί να αυξήσει ε, το κόστος της μεταφοράς και το συνολικό κόστος του προϊόντος. Άλλωστε υπάρχουν και άλλα κριτήρια περιβαλλοντολογικά ε, τα οποία δεν μπορούν να επαληθευτούν σαφώς και δεν μπορούμε να δούμε εάν ένας μειοδότης από τρίτη χώρα ε, ε, παρακάμπτει την νομοθεσία ή όχι εάν προέρχεται από μία συγκεκριμένη χώρα. Ο κύριος Ταραμπέλα δέχεται πλήρως την χαμηλότερη τιμή ενώ θα πρέπει να συγχρόνως ε, να εξασφαλίσει κανείς ε, τις συνθήκες εκτελέσεως της προσφοράς διότι ε, δεν μπορεί για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες το μόνος καθοριστικός παράγωνα είναι η τιμή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία μεθοδολογία μεθοδολογία που θα αποφεύγει τις διακρίσεις. Ενώ αυτό το έχει διαγράψει ο εισηγητές, ο οποίος ζητά να ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως το κοινωνικό κόστο και ε, υπάρχουν ορισμένα σημεία όπως η διαφάνεια η οποία θα έπρεπε να υπολογίζονται πιο πολύ. Οι ε, προϋποθέσεις αυτές ε, τις οποίες καθορίζει ο εισηγητής είναι προβληματικές και μπορεί να αποκλείσει ορισμένους ενδιαφερόμενους από δημόσιους διαγωνισμούς ούτε είναι δυνατόν ε, να ε, ισχύσουν σε νέους διαγωνισμούς προϋποθέσεις παλαιότερων. Ε, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση όλων ενώ ο κύριος Ταραμπέλα ζητά να υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις τις οποίες όμως θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να στηρίξουμε διότι ότι για περίπλοκες ε, περιπτώσεις ενδέχεται να αυξηθεί το κόστος. Ε, γι' αυτό και πρέπει να δούμε ε, πόσο θα λαμβάνουμε τις αποφάσεις. Θα πρέπει σε όλους να δοθούν οι δέουσες δυνατότητες και η χρήση της Διεθνής Συμφωνίας για την ανάθεση των δημοσίων έργων θα πρέπει να ισχύσει με τον κανόνα της αμοιβαιότητος ενώ ο εισηγητής αναφέρεται μόνο στο θέμα της προσβάσεως στην αγορά. Ε, γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να λυθεί ίσως σε άλλες οργανώσεις όπως ο ΠΟΕ. Κύριε Ταραμπέλα, μη μου κρατάτε ε, κακία που αναφέρθηκα σε όλα τα αρνητικά σημεία χωρίς ε, να επενήσω την ε, δέσμευση και την προσπάθειά σας αλλά πρέπει να υπάρξουν και άλλα στοιχεία και αγαπητοί συναδελφοί όπως το είπαμε εχθές πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα συγκεκριμένα να προσέξουμε τις μειώσεις των μισθών διότι ε, δεν ισχύει μόνο το θέμα της διαφάνειας ή στις δημόσιες προμήθειες όπου μπορούμε να συζητήσουμε να ξέρετε ότι θα βρείτε στο πλευρό σας τους φιλελεύθερους.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 και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά επειδή δεν έχουμε επαρκή χρόνο για τροπολογίες και ουσιαστικά δεν θα, θα είναι εκτός μάχης και όλη η εβδομάδα του Στρασβούργου θα έχω μόνο την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένη σήμερα για να μπορέσω να διευκρινίσω ορισμένα θέματα για να μην θέσω άχρηστες τροπολογίες. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση συγκεκριμένα στην πρότασή σας για τον κανόνα των τεχνικών προδιαγραφών που θέλετε να διαγραφεί από το παράθυμα 8 και να μεταφερθεί κάπου αλλού. Θεωρώ ότι είναι καλό να απλοποιούμε αλλά στο τέλος ο κατάλογος επεκτείνεται. Αν αυτή, αυτός ο κατάλογος μεταφέρεται δεξιά και αριστερά, ποιος είναι ο λόγος. Ε, γιατί παραδείγμα το χάρη ε, ε, δεν δέχεστε κατευθείαν ε, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες τα οποία απλούστατα αναφέρονται στο παράρτημα 8. Επίσης τα θέματα των τεχνικών προδιαγραφών διαβίωσης ε, θα έπρεπε να συνεννοηθούμε διότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα έγγραφο ενημέρωση των συντονιστών γιατί είναι πολλά που δεν καταλαβαίνω όπως είπε και η κυρία Βέσλου νομίζω ότι και αυτή συγχαίει ορισμένα πράγματα και αυτό οδηγεί στο ότι διαγράφονται οι διεθνείς προδιαγραφές οι οποίες είναι απαραίτητες εάν θέλω να κάνω μία προκήρυξη και ένα διαγωνισμό σχετικά με το ICT, δηλαδή με τα κομπιούτερ. Ε, οπότε μήπως θα βοηθούσε αυτό το έγγραφο ενημέρωσης να έχουμε μία καλύτερη ε, βάση, να ξέρουμε τι είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και και τι, ε, τι συμβαίνει με τα Third Certified Standards. Αυτό δεν το κατάλαβα, διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για προδιαγραφές, αλλά ε, δεν πρέπει να ε, διαφέρουν οι έννοιες που χρησιμοποιούμε για τους δημόσιους διαγωνισμούς από αυτούς που χρησιμοποιούμε στον καθορισμό των προδιαγραφών, για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις όσον αφορά τη συμφωνία του TBE του Δεκεμβρίου αντιλαμβάνουμε ότι δεν θα ισχύσουν πλέον οι ε, αρχές που είχαν θεσπιστεί. Τότε όμως γιατί δεχτήκατε την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου είπαμε ότι θα πρέπει η παροχή Β να ε, μπορέσει να προχωρήσει διότι ε, μη ένας δήμος που χρειάζεται να στραφεί εναντίον ενός εντολοδόχου χρειάζεται συμβουλή νομική και θα πρέπει να υπάρξει ένας δημόσιος διαγωνισμός πριν αναθέσει τη δουλειά αυτή σε κάποιον. Όταν πρόκειται λοιπόν για διάφορες υπηρεσίες όπως οι συμβολεογράφοι, οι δικηγόροι και ούτω καθεξής θα πρέπει να ισχύσουν εξαιρέσεις τις οποίες δεν έχετε διατηρήσει. Επίσης όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές και τις τιμές κινήσεως. Αυτό το βλέπουμε τον, στην αρμόδια οδηγία σε ένα εκατομμύριο ενώ εσείς αναφέρετε 500.000. Οπότε σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να ε, καλύψει και να προκηρύξει σε ολόκληρη την Ευρώπη διαγωνισμούς για μικρότερα ποσά που μου φαίνεται περιττό και θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε για να δω εάν θα το περιλάβω στις τροπολογίες ή όχι. Για τις υπεργολαβίες το κάλυψαν οι προλαλήσαντες, τα ε, κόστη. Δεν θέλουμε να πάρουμε τον απόλυτο μειοδότη, αλλά από την άλλη πλευρά για διάφορα ε, τυποποιημένα προϊόντα θα αποφασίσουμε βάσει της τιμής. Εάν λοιπόν κατάλαβα σωστά αυτά τα οποία είπατε και περιγράψατε, ε, είπατε ότι είναι υποχρεωτικό να δεχθεί κανείς ε, την πιο ενδιαφέρουσα προσφορά χωρίς να λάβουμε υπόψη την τιμή, πράγμα το οποίο θα είναι προβληματικό γιατί δεν μπορεί να ισχύσει παντού. Σε ορισμένα προϊόντα θα πρέπει να αποφασίσουμε βάσει της τιμής αλλά να συμφωνήσουμε ότι θα είναι περιορισμένα προϊόντα και εκεί θα ισχύσει η πλέον ε, οικονομική προσφορά. Εν ολίγης, δεν καταλαβαίνω πώς οι δομές αυτές θα ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να περιγραφούν, διότι στη Γερμανία παραδείγματο χάρη υπάρχουν ομοσπονδιακές δομές. Εσείς ε, αλλάξατε το άρθρο 54, θα υπάρχουν ε, προβλήματα και θέλω να υπάρξει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια με την αναθεώρηση και όχι ασάφεια και περισσότερα προβλήματα σχετικά με την τροπολογία 86 και 87 όπου λέτε ότι αρχικά ε, υπάρχει το θέμα της χρησιμοποίησεως των συλλογικών συμβάσεων και εκεί ε, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη κάτι τέτοιο πρέπει να δώσουμε τον ακριβή ορισμό. Επίσης ε, είπατε σε κάποιο σημείο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο προστασίας και να αποφύγουμε τις, τους αποκλισμούς. Αλλά εάν δεν διευκρινίσουμε ακριβώς τι εννοούμε εδώ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε σταφείς, θα υπάρξουν ε, πολλές, ε, πολλά προβλήματα και πρέπει να υπάρχουν πιο σαφείς ορισμοί. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, κάνατε μια πλήρη τοποθέτηση. Κυρία Ρούλα, δεν με ακούτε. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούσα για την καθολική άποψη που καταθέσατε. Και θέλω να υπενθυμίσω και την προηγούμενη δουλειά σας ε, ως εισηγήτρια που οδήγησε προς αυτή την ε, πρόταση, ο κύριος ε, Κόζουσνικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν αρχίσαμε να εργαζόμαστε επί των δημοσίων συμβάσεων, συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στους μελλοντικού διαγωνισμούς, ε, προσβάσιμε στις μέσες επιχειρήσεις, να είναι πιο διαφανή και να είναι και πιο εύκολη διαδικασία για τι αναθέτουσε αρχέ. Όταν ε, βλέπω την πρόταση που έχουμε ενώπιόν μα, Όταν είδα την πρόταση, θυμήθηκα μία δήλωση ενός ε, πολιτικού από το παρελθόν. Ίσως θα μπορούσαμε εδώ να κάνουμε ένα διαγωνισμό για να δούμε ποιος θα το γνωρίζει. Και το άτομο αυτό ήθελε την αλλαγή, ήθελε τη βελτίωση, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ε, το συνηθισμένο. Εμένα μου αρέσει το τμήμα που αφορά τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να έχει πάει και πιο μακριά εισάγοντας ε, μια τυποποιημένη διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού, κάτι που θα ήταν πιο διαφανές ε, και που θα μπορούσε να εφαρμόζεται και σε εθνικό επίπεδο. Όμως ε, εγώ νομίζω ότι εδώ παρασυρθήκαμε κάπως από τις ουτοπίες. Χαίρομαι που σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Γιούρη Νομικών Θεμάτων όπου είχαμε και εκπροσώπους ε, από διάφορους τομείς. Συζητήθηκαν ακριβώς αυτά τα κριτήρια, τα κοινωνικά και μάλιστα και κάποιος εκπρόσωπος ε, από τη Σουηδία μίλησε ε, για το θέμα αυτό και τοποθετήθηκαν και τα συνδικάτα σχετικά. Εγώ νομίζω πάντως ότι αυτές οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κυρίως όταν έχουμε χαμηλές τιμές αλλά και επίση όταν και οι κοινωνικές ε, συνθήκες και ισότητα των ευκαιριών λαμβάνονται υπόψη γιατί διαφορετικά οδεύουμε προς την κόλαση. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε κατά νου ότι με αυτή την νομοθεσία αν ε, δεν νομοθετήσουμε σωστά, τότε θα εξάγουμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου την οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μιλάμε για πραγματική τραγωδία. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και αυτά τα δικαιώματα. Το είπε και ο Γιώργο Κρόιτσμαν. Εξακολουθούμε να έχουμε χρόνο για άλλα, να αλλάξουμε αυτή την νομοθετική πράξη. Έτσι λοιπόν α αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εφιαλτική κατά κάποιο τρόπο συνεισφορά σας. Είναι ένας τομέας που όλοι πρέπει να εξετάσουμε. Ο κύριος De Jong είναι ο τελευταίος ε, ομιλητής ε, και όταν το ολοκληρώσει ο κύριος De Jong ε, να ελέγξω, έχω 8 άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Αν κάποιο άλλο θέλει το λόγο, τώρα να μα το γνωστοποιήσει, γιατί πρέπει να σεβαστούμε και το χρόνο. Να σα πω ποιοι είναι στον κατάλογο μετά τον κύριο Διόγκ. Mr. Mrs. Uh, Mrs. corazza Άλλος κανείς? Και κύριε Πετικάινεν, ε, νομίζω ότι νωρίτερα είχατε στήσει το λόγο. Μάλιστα θα αφαιρέσω τον πρώτο πρόεδρε από τον κατάλογο. Κάποιος άλλος? Όχι. Λοιπόν, αφού θα μιλήσει ο κύριος Ντογιόγκ, Θα προσπαθήσουμε να μην μακρηγορήσουμε για να μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο και να μπορέσει να συνεισφέρει και η Κομισιόν. Κύριε Ντεγιόνγκ, από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά αυτή τη φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάρκα Ταραμπέλα για την εκθεσή του. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά σημεία σε αυτό το σχέδιο κειμένου. Σε σχέση με όσα είπαν ε, και οι προηγούμενοι ομιλητές για τα κοινωνικά κριτήρια, θέλω να πω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Μιλήσαμε στο παρελθόν ε, για συμβάσεις ε, καθαριότητας και Νομίζω ότι, παραδείγματο χάρη, ε, εγώ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μια τουαλέτα που καθαρίζεται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Βλέπετε λοιπόν ε, ότι υπάρχει και μια δυσαναλογία μεταξύ της, μια αναλογία με της, ε, μεταξύ της υπηρεσίας που παρέχεται και των εργα εργασιακών συνθήκων. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, δεν θέλουμε μόνο καθαρέ τουαλέτε, αλλά θέλουμε να έχει και αξιοπρεπή εργασία το προσωπικό. Έτσι λοιπόν, ε, κυρία Ταραμπέλα, δράτε την ευκαιρία για να το θέσουμε αυτό στην ημερησία διάταξη και βλέπουμε σε όλα τα θέματα να αν μην αναφέρονται τα κοινωνικά ζητήματα, όμως ε, πραγματικά εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα πράγματα στα οποία συζητούμε. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της έκθεσης και θα ήθελα να το υπερασπίσουμε εμείς ε, με ισχύ σε αυτή την Επιτροπή. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία από τη δική μου ομάδα. Νομίζω ότι μπορούμε να αυξήσουμε αυτό το κατώτατο όριο Μιλάμε για εταιρείε ε, που δεν δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλές εταιρείε δεν δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί δεν ξέρουν ποιε είναι οι απαιτήσει. Ε, όχι επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγες μειοδοτικές ε, διαδικασίες στην Ευρώπη. Υπάρχουν οι υπηρεσίες πανευρωπαϊκές και μπορούν να υπάρξουν ε, τέτοιες συμβάσεις, αλλά ξέρετε ε, υπάρχει δυσκολία σε σχέση με τα κατόφλια. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα έπρεπε να ρεύουν τα κατόφλια αυτά και σε σχέση με την οντότητα, οντότητα ελέγχου. Εδώ θα ήμουν κάπως προσεκτικός σε σχέση με τη σύσταση νέων φορέων. Ο κ. Τεραμπελή είπε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους φορείς Όμω αυτή η παρακολουθήση ήδη γίνεται, γίνεται ήδη από τι τοπικές αρχές και αναρωτιέμαι αν θα χρειαζόμαστε μια ξεχωριστή οντότητα παρακολούθησης ε, της ε, διαδικασίας του διαγωνισμού. Θα πρέπει να με πείσετε για το θέμα αυτό. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω, νομίζω ότι είναι ζωτική σημασίας, κάτι που θα πρέπει να είναι το σημείο εστίασης ότι οι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο. Νομίζω ότι η Κομισιόν βρίσκεται στη σωστή οδό και το ανέφερε και ο κύριο Ταραμπέλα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Α προχωρήσουμε λοιπόν στου ευρωβουλευτέ. Κύριε Βάις Κέμπερ, πρέπει να φύγει σε 20 λεπτά. Έτσι λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα προλάβει να πάρει το λόγο. Εννέα άτομα έχουν ζητήσει το λόγο και έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Έτσι λοιπόν θα σας παρακολούσα να περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Και μετά να ακούσουμε και την Κομισιόν. Ξέχασα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Όμως ε, ξέρω ότι σήμερα το απόγευμα είναι και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και υπάρχει και κάποιο feedback από την πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω η κυρία Νιέτη είναι εδώ από την Κομισιόν και θα απαντήσει τις ερωτήσεις. Έτσι λοιπόν, ε, δύο λεπτά να σας δώσω ενδεικτικά και να ακολουθήσουμε την εξή σειρά. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Πετικάινεν, πιστεύω, που ζήτησε το λόγο νωρίτερα και κατόπιν να ακούσουμε την κυρία Στόιλε, την κυρία Βάισκεβερ, την κυρία Χάντσλι και τον κύριο Τζουρβά, την κυρία Κορατσαμπίλ και τον κύριο Κορφεράτη Κυρία Γκέπαρτ, είστε όλοι ικανοποιημένοι. Ε, αν κάποιο άλλο θέλει το λόγο πριν από μένα, ευχαρίστω. Όχι, όχι, εσεί νομίζω πρέπει να πάρετε το λόγο πρώτοι. Ε, Αρκεί να μιλήσουμε όλοι για δύο λεπτά. Έχετε το λόγο ω πρώτη αντιπρόεδρο για δύο λεπτά. Και εγώ θα ξεγλιστρήσω για να δω τους βουλευτές από την Ιαπωνία. Ξέρω ότι σας αναφέρω δύσκολη δουλειά εδώ να προεδρεύσετε σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να θίξω ορισμένα από τα ζητήματα για να είμαστε κάποιο πιο επικοδημητικοί. Καταρχήν, στρατηγική για τις δημοσίες συμβάσεις. Νομίζω πρέπει να αλλάξουμε όλη τη σειρά για το πώ υλοποιούμε τι δημοσίε συμβάσει. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια πολιτική διαδικασία όπου ε, εξετάζουμε όλα τα κριτήρια, δηλαδή να έχουμε μια πολιτική συζήτηση τι θέλουμε από το προϊόν, από την υπηρεσία που παρέχεται, παραδείγματο χάρη ε, για τους ηλικιωμένου ή για τους μαθητές το σχολείο και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό να έχουμε μια δημόσια ακρόαση αν ε, αυτές οι υπηρεσίες αφορούν ε, ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως το χάρη η παροχή τροφίμων στα σχολεία, ή υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους. Θα έπρεπε λοιπόν να είναι υποχρεωτικό να υπάρξει μια κρόση και να ακούσουμε όσους χρησιμοποιούν και αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, ε, τώρα γίνεται το αντίστροφο. Πρώτα έχουμε το μεδοτικό διαγωνισμό και κατόπιν έχουμε την πολιτική διαδικασία. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα τώρα για τι ηλεκτρονικέ δημόσιες συμβάσει. Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να προχωρήσουμε με τολμηρά βήματα. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να έχουμε ε, μία, ένα ομοιόμορφο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας που θα μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες και έτσι θα βοηθούσαμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να βρουν τις προσφορές. Αυτό θα διευκόλυνε και τους μειοδότες όσους υποβάλλουν τις προσφορές ε, και θα αποφεύγαμε και διάφορα λάθη. Παραδείγματο χάρη να γίνονται προσφορές μόνο βάσει τιμής. Κατόπιν, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Η... Αυτό το θέμα χρειάζεται να το σκεφτούμε. Επίσης, ε, θα πρέπει να γίνεται και υποχρεωτική ανάλυση του κύκλου της ζωής ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και θα πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξο ποσοστό περιβαλλοντικό ε, για όλες ε, τις δημόσιες συμβάσεις. Τώρα τα ελάχιστα κριτήρια για όλους ε, θα πρέπει να είναι να σέβονται τους κανονισμούς της ΔΟΕ και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για ε, τις συνθήκες εργασίας και για τη δημόσια φορολογία. Γιατί δεν θέλουμε να ζημιώσουμε τους εαυτούς μας και τις αγορές μας με εταιρείε που δεν σέβονται τα κριτήρια, τους κανόνες. Πρέπει να ολοκληρώσω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ε, κοινή ευθύνη, ε, πρέπει να δούμε τι κάνουν οι επιχειρήσει με τι συμβάσει, τι βάζουν στι συμβάσει και σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση τη καινοτομία. Νέε μέθοδοι πέρα από τα τεχνικά κριτήρια θα πρέπει να αποτελούν ε, ένα παράθυρο για τους μελλοντικού διαγωνισμού βάσει αποτελεσμάτων. Δηλαδή, να βλέπουμε τι θέλουμε να πετύχουμε με την ίδια τη διαδικασία. Παραδείγματο χάρη, χρειάζομαι αυτά τα δύο έγγραφα να είναι μαζί, αντί να ζητήσω συνδετήρε. Και έτσι προωθούμε την καινοτομία. Λυπάμαι, αλλά προσπαθήστε να μην ξεπερνάτε το χρόνο των δύο λεπτών, γιατί αν μιλάτε όλοι τρία και τρισήμιση λεπτά δεν θα καταφέρουμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τον εισηγητή πάλι στο τέλος. Κυρία Μπέισμπεργκ, εφόσον πρέπει να φύγετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την κατανόηση γιατί θα ήθελα να προλάβω το αεροπλάνο μου. Καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρόστασή του και θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής. Καταρχήν ε, συμφωνώ διότι χρειαζόμαστε και κοινωνικά κριτήρια και περιβαλλοντολογικές σκοπιμότητες αλλά και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά θα ήθελα αυτό να είναι ε, εθελοντικό διότι πολύ σωστά ε, το είπε και η κυρία Ρούλε η υποχρέωση είναι υπερβολική και θέλουμε να διευκολύνουμε τις διαδικασίες διαδικασίες, να τις καταστήσουμε πιο ευέλικτες και αυτό είναι αντίθετο με μία υποχρέωση, χωρίς να είμαστε αντίθετοι. Θέλουμε απλώς να είναι κάτι εθελοντικό. Όσον αφορά το ο κριτήριο της ε, προσθήκης θεωρώ την πρόταση του ομιλητή ενδιαφέρουσα και ε, η τιμή είναι ένα θέμα αυτής της, ε, αυτής της αξιολόγησης αλλά δεν χρειάζεται να είναι τόσο ασαφές. Ε, επίσης ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εάν ε, θα περιοριστούν οι διευκρινήσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι και καθορισμένες χρονικά και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να διευρυθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια για να μπορεί ε, να ε, συντονίσει την ε, προσφορά με τις ανάγκες. Πέραν αυτού, όσον αφορά τις τιμές εκκινήσεως, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ χαμηλές αυτές τις οποίες ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να αυξηθούν, διότι δεν ανταποκρίνονται εις την αγορά έτσι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ζητώ λοιπόν μία αύξηση των ε, κατοτάτων τιμών ε, και όσον αφορά την υπεργολαβία και την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να προσέξουμε να μην συνδυάσουμε πάρα πολλές ε, υποχρεώσεις και να προσθέσουμε και την εποπτεία που θα βαρύνουν πολύ το μηχανισμό. Ε, πιστεύω ότι όσον αφορά την governance ε, είμαι αρνητική γιατί δεν θέλουμε να ενισχύσουμε τη γραφειοκρατία Δημοκρατία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Ζουβά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεδομένη της πολυπλοκότητας του κειμένου μπορούμε να συμφωνήσουμε ή όχι σε κάποια σημεία με τον εισηγητή, αλλά από αντικειμενικής πλευράς, και αληθεύει εδώ πέρα αυτή τη φορά, έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερον, δεν έχω πολύ χρόνο στη θέσή μου, δεν μπορώ λοιπόν να μιλήσω για όλα αυτά τα θετικά που βρίσκω στο κείμενο. Θα επικεντρωθώ στα αρνητικά σημεία και σα ζητώ συγγνώμη κύριε Ταραμπέλα. Όταν λέω αρνητικά, ενώ ουσιαστικά ότι χρειάζομαι περισσότερε εξηγήσει για κάποια σημεία. Καταρχά, πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε προ διαδικασίε πιο ευέλικτε και θα πρέπει να ευνοήσουμε περισσότερο και να καταστήσουμε πιο εύκολη την εργασία που κάνουν οι εθνικές αρχές. Ενδεχομένως να πρέπει να γενικευθούν και οι ε, διαδικασίες ε, διαπραγμάτευσης με ανταγωνισμό. Οι προτάσεις που κάνει ο εισηγητή, νομίζω ότι πολλέ φορέ μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια αντιφατικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι τροπολογίε που καταργούν την μείωση τη προθεσμία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά στερούν από το δημόσιο τις δυνατότητες που του δίναμε στην αρχική μας πρόταση. Επίσης, οι κανόνες που έχουν να κάνουν με την ανάθεση όπου περιορίζονται τα κριτήρια ουσιαστικά πάλι βαίνουν κατά του δημοσίου, των δημοσίων αρχών που θα έπρεπε ουσιαστικά να έχει το δημόσιο, δημόσιες αρχές, το εργαλείο αυτό που του είχε δώσει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης κάποιες τροπολογίες όπως 127-128 για που προβλέπεται ένα πολύ χαμηλό κατόφλι. Νομίζω ότι το κατόφλι αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν μπορεί να γίνει κατάλληλη αξιολόγηση μέσω των χαμηλών αυτών τιμών. Σαφώς θα πρέπει να θέσουμε κάποιες κυρώσεις κατά των πολύ χαμηλών τιμών, αλλά με τις τροπολογίες που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κατάλληλη αξιολόγηση της προσφοράς. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες ε, παραδόξως ε, είναι κατά των δημοσίων αρχών, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούνται εδώ πέρα κάποια κριτήρια τα οποία επιβάλλουν συγκεκριμένε υποχρεώσεις. Και το ρήμα «may» αντικαθίσταται από το «σαλ» και θεωρώ όμω ότι καταλήγουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Θα προσθέσω επίσης κάποιες ακόμα παρατηρήσεις και ολοκληρώνω δεν καταφέρνω τελικά να αποφασίσω για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τη διάκριση των υπηρεσιών προτεραιότητας και μη προτεραιότητας. Καταργώντας τη διάκριση αυτή, μήπως τελικά περιορίζεται τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να έχανε μια πιο ελαφριά διαδικασία προσφοράς και ανάθεσης και μήπως πετυχαίνετε πάλι το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο θέλετε να πετύχετε στην αρχή. Και τέλος, ε, οι ψηφιακέ ε, υπηρεσίε, Ναι, σαφώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προ την ψηφιοποίηση αυτή. Μήπως όμως να περιορίσουμε την υποχρέωση αυτή προ ε, τις δημόσιες αρχές, αλλά από την άλλη οι άλλοι φορεί, οι ιδιωτικοί φορεί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ενδεχομένω να μην πρέπει να περιορίζουν, να μην πρέπει να βαρύνονται από αυτή την υποχρέωση της χρησιμοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών. Μάλιστα, από ό,τι κατανοώ είναι πολύ πλοκοτό θέμα και δύσκολο και κανένα δεν μπορεί να περιοριστεί στα δύο λεπτά. Ο κύριος Κομφεράτη τώρα. Μετά. Μετά εσείς. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο. Σε ό,τι αφορά δύο σημεία που φαίνονται κεντρικά για το θέμα, δηλαδή το κατόφλι ε, το ελάχιστο που αποτελεί καταστροφή σε πάρα πολλέ χώρε ε, στο να περάσουμε στην πλέον συμφέρουσα οικονομικό προσφορά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό και κυρίω και αυτό ίδιο ισχύει ό,τι αφορά και την υπεργολαβία. Στην δική μου χώρα υπάρχει πολύ περιοριστική νομοθεσία για το θέμα αυτό και οι περιορισμοί αυτοί παρόλα αυτά δεν έχουν ποινικοποίησει τις επιχειρήσεις, ούτε σκότωσαν κανένα, αλλά μάλιστα ε, δυστυχώς ε, διαιωνίζεται η παρουσία των ε, κακοποιών, γιατί κυρίως εκεί όπου έχουμε πολύ ε, αστηρούς διαγωνισμούς έχουμε, ε, ευνοείται μάλλον η παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος και θα ήθελα να σταθώ σε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά τις μικρές ε, και μεσές επιχειρήσεις. Εγώ δεν συμφωνώ με το ότι για να βοηθήσουμε τις μεσές επιχειρήσεις θα πρέπει να κατακαιρματίσουμε τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Είναι δύσκολο να τους κατακαιρματίσουμε τους διαγωνισμούς και ο κατακαιρματισμός μπορεί να γίνει κάτι αυθαίρετο, χωρίς αιτιολογία και, και αυτό να σημαίνει ότι ποινικοποιούνται οικονομικά και οι ίδιες επιχειρήσεις. Αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι γιατί θα πρέπει να δώσουμε κίνητρο να ενοποιούνται οι μικρέ επιχειρήσει για να συμμετέχουν στου διαγωνισμού και να δίνουμε τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσει για να γίνουν μεγάλε και να εργαζόμαστε σε συντονία με άλλα παρόμοια υποκείμενα χρησιμοποιώντα τι συνέργειε που θα μπορούσαν να υπάρξουν ε, μεταξύ ε, συναφών αλλά όχι ταυτόσιμων δραστηριοτήτων. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τι αντικειμενικέ συνθήκε που υπάρχουν σε κάποιου τομεί. Έχουμε δημόσιου τομεί ε, που τίθενται υποδιωτικοποίηση. Πολλές φορές είναι μακροσκελή η διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι για τι επιχειρήσει που βρίσκονται μέσα σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίηση ε, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ειδικό καθεστώ. Δεν με πείθει η ιδέα να ε, αφαιρέσουμε όλο τον τομέα από την ε, διαδικασία που καθορίζουμε, γιατί διαφέρουν και συνθήκε από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπερισχύσει η αρχή τη μη ποινικοποίηση, δηλαδή τη ομοιομορφία στι συνθήκε. Όμως αυτές οι συνθήκες ε, θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι ε, δυνατόν να τεθούν ε, σε πράξη σε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ θα περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο. Αυτό και για να αποφύγουμε κάποιες διαδικασίες ανταγωνισμού στο ερικό της ίδιας χώρας συνήθως και όταν μιλάμε για μονοπόλιο, για να αποφύγουμε διαδικασίες που αλλοιώνουν τις δυναμικές της αγοράς μεταξύ διάφορων χωρών, από χώρα σε χώρα. Η κυρία Χανσλίκ έχει τώρα το λόγο, δεν σας έχω ξεχάσει. Ε, <laughs> Ευχαριστώ. Χαίρομαι που δεν με ξεχάσατε. Δεν ξέρω αν ε, μπορώ να σεβαστώ το χρόνο, τα τρία λεπτά που μας έχετε δώσει. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τεραμπέλα για την εξαιρετική δουλειά του. Ξέρω ότι δύο λεπτά θα έπρεπε να έχουμε κανονικά, αλλά κοιτάξτε, όλοι τρία μίλησαν. Τώρα, για να επανέλθω στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων σε δύο πολύ σημαντικές ε, πτυχές. Ε, καταρχήν, αυτές οι λεγόμενες ε, reserved contracts, αυτές τις συμβάσεις Ξέρετε ότι η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη ε, και το τι γίνεται με ανθρώπους που είναι σε μειονεκτική θέση. Τώρα όμως έχουμε απελευθέρωση αυτές τις ρήτρες, έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι για τις κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιβαίνουμε στη συνθήκη κυρίως ό,τι αφορά τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ο κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι καταρχήν να καταστήσουμε πιο ευέλικτε τις διαδικασίες και να υπάρχει καλύτερο streamlining και νομίζω ότι οι στόχοι των άλλων πολιτικών θα πρέπει να συνάδουν και με αυτούς εδώ τους στόχους. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, όμως ε, δεν μπορούμε να μπερδεύουμε αυτά τα δύο θέματα με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Δεύτερο ζήτημα. Διαπραγματεύσεις χωρίς πρώτερη προκήρυξη. Αναφέρομαι στο άρθρο 30. Εδώ έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα. Καταρχήν, το opting out, ε, δηλαδή ε, opting out για τις δημόσιες συμβάσεις που είναι ε, δευτερογενείους φύσεως. Όταν μιλάμε για μια μεγάλη σύμβαση και πρέπει να συμπληρωθεί με μια δευτερογενή διαδικασία, γιατί δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε τα πάντα εξ αρχής, αυτό πρέπει να το λέβουμε υπόψη. Και δεύτερον, αν συγκρίνουμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή στο κανονισμούς, στους κανονισμούς, Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που ορισμένες συμβάσεις ε, δεν μπορούν να τεθούν για καλλιτεχνικούς λόγους. Ε, Παραδείγματο χάρη, ε, μιλώ για την αγορά έργων τέχνης, αλλά μπορεί να ληφθούν υπόψη και άλλοι λόγοι καλλιτεχνικής φύσεως. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για ένα έργο τέχνης αυτό καθ' αυτό. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτες όταν έχουμε να κάνουμε με συμβάσεις που έχουν κάποια συγκεκριμένα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά. Και τελευταίο σχόλιο, η διαδοχική υπεργολαβία αναφέρομαι στο άρθρο 34 ρήτρα 3. Τρία, δεν θα ήταν αντιπαραγωγικό, δεν θα μας οδηγούσε αυτό στον αποκλεισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και τελευταίο θέμα, ε, έχουμε και το τομεακή οδηγία, δεν το συζητήσαμε αυτό, αλλά είναι σημαντικό. Σε ορισμένου τομεί έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένε συμβάσει στι ταχυδρομικέ υπηρεσίε. Παραδείγματο χάρη, έχουμε απελευθερώσει εντελώ τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε. Θα ήταν λοιπόν απαραίτητο να καλύψουμε και αυτόν τον τομέα που βασικά υπάρχει βάση, στον ελευθερο... βάση του ελεύθερου Σα ευχαριστώ και σα ευχαριστώ για την υπομονή σα. Ευχαριστούμε, κυρία Στάιλερ. Στήλερ. Στήλερ, συγγνώμη. Στάιλερ. Πολύ γρήγορα, ούτε ένα λεπτό δεν θα χρησιμοποιήσω. Θα ήθελα να γνωρίσω περισσότερα πράγματα όσον αφορά τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Bon. Merci. Ευχαριστούμε. Κοράτσα Μπίλτ. Μπορώ να πάρω βέβαια το χρόνο της Κάθριν. Πολύ ευχαρίστως. Τρεις ομιλητές έχουμε ακόμα στον κατάλογο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον πρόεδρο που καλωσόρισε την ομάδα επισκεπτών από τη Σουηδία. Να πω στον Μάρκ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι επικεντρώνεται σε δίκαιους, απλούς και ευέλικτους κανόνες. Αλλά στο κείμενο τι βλέπουμε μετά, ότι προσθέτουμε κριτήρια, προσθέτουμε συνθήκες και τελικά καταλήγουμε να είμαστε ασαφείς. Ας είμαστε λοιπόν πιο συνεπείς. Τέσσερα σημεία. Συμφωνώ με τον κύριο Ρούλερ. Συλλογικές συμβάσεις. Ποια είναι η σχέση τέλο πάντων με το κείμενο αυτή τη στιγμή μία μέθοδος βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε κανόνες εσωτερικής αγοράς. Εδώ πέρα μιλάμε για δημόσιες συμβάσεις και θα πρέπει να καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε πώς λειτουργούν ή πώς θα λειτουργήσουν οι χιλιάδες αυτές δημόσιες αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσουν το κείμενο αυτό προκειμένου με δημόσιους πόρους να χρησιμοποιήσουν, να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Η σαφήνεια. Η σαφήνεια είναι ο καλύτερος τρόπος που θα οδηγήσει τελικά σε ευελιξία τόσο να αφορά τα συστήματα ελέγχου και το σύστημα υπεργολαβίας. Θεωρώ ότι και εδώ πέρα δημιουργούμε επιπρόσθετη γραφειοκρατία που δεν θα πρέπει να έχει καμία θέση στο κείμενο αυτό. Η βασική μου ανησυχία έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Τρόφιμα για τα παιδιά, τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους, όπως είπατε κι εσείς, τους παθητικούς λεγόμενους καταναλωτές που θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα σε ποιοτική υγιεινή διατροφή όπως οποιοδήποτε άλλος. Και έπειτα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όχι μόνο την πιο φτηνή επιλογή, αλλά την επιλογή εκείνη που δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων για τα τρόφιμα μπορεί τελικά όντως να δώσει πρόσβαση στους μικρότερους παράγοντες στην αγορά και επίσης μπορεί να μας βοηθήσει να αποκριθούμε στην πολύ μεγάλη ζήτηση που υπάρχει από τους Ευρωπαίους πολίτες για φρέσκα εποχικά προϊόντα τα οποία παράγονται με φιλικούς προς το περιβάλλον ε, τρόπους που δεν, δεν συμβάλλουν στις κλιματικές αλλαγές και δεν ζημιώνουν το περιβάλλον. Τροπολογία 34 τώρα. Κύριε ε, Μάρκ, τι εννοείς όταν λες η τοποθεσία της παραγωγής να αποτελεί κριτήριο. Μα μιλάμε αυτή τη στιγμή για έναν για μια νομοθεσία εσωτερικής αγοράς όπου δεν θα πρέπει να δημιουργήσει καμία περίπτωση διακρίσης. Βλέπω ότι η διατύπωση που χρησιμοποιείται εδώ πέρα ενδεχομένω να οδηγήσει σε προβλήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Βάιλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα περιοριστώ σε τρία σημεία. Το ένα είναι ότι διαπίστωσα ότι γίνεται μία συζήτηση τώρα και ασχέτως της ε, ε, της κομματικής μας τοποθετήσεως θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να υπάρξει πράγμα το οποίο δεν ίσχυε στην προηγούμενη εξέταση προεφτά ετίας. Επίσης θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ε, και δεν μπορούμε μπορούμε να λέμε ότι ε, πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν ξέρουν τι κάνουν διότι οι ε, εταιρείε οι οποίες ε, αναλαμβάνουν διαγωνισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να σεβαστούν τις συλλογικέ συμβάσεις. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτές, άρα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σε όλες τις χώρες και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο. Επίσης ε, η αποκαλυπτική θεώρηση μου φάνηκε ότι δεν ήταν σωστή. Βέβαια ήταν ε, πολύ συγκινησιακή αλλά ε, υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες από την κεντρική Ευρώπη τους οποίους εκμεταλλεύονται στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Οπότε θα σας παρακαλώ να μην ε, ε, ε, χρησιμοποιείτε ορισμένα σοσιαλιστικά οράματα που δεν μας οδηγούν πουθενά. Αλλά το παράδειγμα το οποίο αναφέρατε για τις καθαρίστρες και τους καθαριστές που έχουν όλο και μεγαλύτερη πίεση αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιληθεί ε, στο επίπεδο όπου ρυθμίζονται οι συλλογικέ συμβάσει. Δεν επιπλήττω εσάς, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, το θέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή ε, πρέπει να πληρώνουν αυτές τις γυναίκες κάτι παραπάνω ακόμη και εάν πληρώνει περισσότερα ο καταναλωτής και φορολογούμενος. Θεωρώ όμως ότι ο τομέας αυτός είναι πολύ ε, περίπλοκος, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλο το θέμα και παρακαλώ ειλικρινά τους ε, συντονιστές, τον εισηγητή, τους κοιόδης να ξανασκεφτούν μήπως θα ήταν δυνατόν τουλάχιστον Λοιπόν, ε, να παρατείνουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες κατά δύο-τρεις εβδομάδες. Λαμβάνετε υπόψη το ζήτημα, θα το εξετάσουμε. Κύριε Ευχαριστώ. Σχετικά με το τελευταίο θέμα θα το ξανασυζητήσω με τον εισηγητή γιατί ενδεχομένως όντως αξίζει να το ξανα Έχω όμως τρία θέματα τα οποία, δεν, ε, στα οποία θα περιοριστώ γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Καταρχήν τα κριτήρια επιλογής και πώς τα αντιμετωπίζουμε και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα για την εξαιρετική εργασία την οποία έκανε και θέλω να υπενθυμίσω ότι τα κοινωνικά κριτήρια έχουν συμπεριληφθεί και στο ισχύον δίκαιο, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι θέλει να διευκρινίσει ορισμένα θέματα και αυτό δεν με ενοχλεί, αλλά δεν πρέπει στο να ε, ε, καταστήσει κανείς πιο συγκεκριμένα να περιορίσει ορισμένα δικαιώματα όπως είναι η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ούτω καθεξής. Να μην λέμε ότι επινοήσαμε κάτι νέο αλλά να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι ε, διατυπωθεί θα είναι σωστό με αποτελεσματικά κριτήρια και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσχυε μέχρι τούδε στο δίκαιο αυτό το οποίο οικονομικά είναι πιο συμφέρον και όχι το φθηνότερο τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε ε, την, ε, τον οικονομική παράμετρο σε σχέση με άλλα θέματα ενώ πρέπει να συνυπολογίσουμε τις κοινωνικές πτυχές την ε, σοβαρότητα ε, των, ε, της εκτελέσεως των παραγγελίων και την βιωσιμότητα διότι στη Γερμανία ίσως η κατάσταση διαφέρει από αλλού όπου υπάρχουν μεγάλες, μεγάλοι διαγωνισμοί κανείς δεν ε, παραμένει στην προσφορά αλλά τελικά πληρώνεις 10, 20, 30 μέχρι και 40% περισσότερο από ό,τι είχε προϋπολογιστεί. Άρα για μένα αυτό που είναι πιο βασικό είναι η ποιότητα και όχι τόσο η χαμηλή τιμή. Και το τρίτο ε, η υπεργολάβη. Βεβαίως θα πρέπει τα κριτήρια επιλογής τα οποία χρησιμοποιούμε για τις προκηρύξεις να ισχύουν και για τους υπεργολάβους γιατί πολλές φορές οι πρώτες επιχειρήσεις τα αναλάβουν και εάν θέλουμε να σεβαστούν τις συλλογικέ συμβάσεις ε, στο υψηλότερο επίπεδο αλλά μετά δεν εφαρμόζονται στους υπεργολάβους τότε δεν κερδίζουμε τίποτα. Όλοι θα πρέπει πρέπει να συμπεριληφθούν και να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και αυτό το σημείο για μένα ήταν πολύ βασικό. Μάλιστα, το λόγο έχει εκπρόσωπος της Κομισιόν για να αντιδράσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ε, είδαμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του κυρίου Τεραμπέλα. Θα είμαι πολύ σύντομη και θα επικεντρωθώ σε τέσσερα σημεία. Καταρχήν, ως ε, Κομισιόν και καθώς περιβρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το τι μπορεί να είναι επιζήμιο για την εσωτερική αγορά. έννοιε όπω η τοποθεσία της παραγωγής είναι κάτι πολύ ανησυχητικό από τη κοπιά της Κομισιόν τουλάχιστον. Και επίσης οι εκκλήσει που άκουσα σήμερα σχετικά με το να αυξηθεί το κατόφλι να αυξηθούν το κατόφλι, να είστε προσεκτικοί στο φαινόμενο κατακαιρματισμού της εσωτερικής αγοράς και επίσης η διάκριση α και β. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτή τη διάκριση και αν ε, σέβεστε την εσωτερική αγορά πρέπει να γνωρίζετε ότι στον κατάλογο Β έχουμε υπηρεσίες με πάρα πολύ υψηλό διασυνοριακό ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν η πρόθεση της Κομισιόν είναι πράγματι να διευρύνει το διασυνοριακό ανταγωνισμό. Το δεύτερο σχόλιο μου έχει να κάνει με κάτι που ήδη υπόθηκε. Να είστε προσεκτικοί ε, με την οριστία, γιατί η οριστία είναι αντίθετη στην ασφαλεία δικαίου και αντίθετη στην απλούστευση και ένας από τους μεγάλους μας στόχους ε, στην εκπόνηση της πρότασης ήταν αυτός να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα νομικά προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη ασφαλής δικαίου και να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερους κανόνες που μπορούν να εφαρμοστούν πιο καλά. Έτσι λοιπόν η οριστία είναι μια ανοιχτή πόρτα ε, για να αυξήσει την προσφυγή στα δικαστήρια και να αυξήσει τις δυσκολίες ε, των αναθεψών αρχών να εφαρμόσουν τους κανόνες. Κάτι ακόμη σε σχέση με την αύξηση της γραφειοκρατίας και για τις αναθέτουσες αρχές και για τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ένα τέταρτο σημείο αμοιβαιότητα. Να είστε προσεκτικοί. Να μην μπερδεύετε τις έννοιες αυτές. Έχουμε μία πρόταση της Κομισιόν για ρύθμιση του θέματος αυτού για ένα κανονισμό και δεν είναι το κατάλληλο θέμα να ρυθμιστούν τα θέματα αυτά σε μια οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτά ήθελα να πω, αλλά βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση ενδεχομένως έχετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος εισηγητής ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές σημειώσει και θα προσπαθήσει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ναι. Ενδεχομένως να απογοητεύσω όμως κάποιους συναδέλφους, αγαπητή Μπερναντέτε, γιατί έχω κρατήσει 7 σελίδες σημειώσεις. Θα προσπαθήσω πάντως να αναφερθώ περισσότερο σε ερωτήσεις οι οποίες ακούστηκαν περισσότερο. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Βάντεν Κάπα από το ΕΛΚΑ, ο οποίος μίλησε εξ του συγητή. Κοιτάξτε, όντως σε σχέση με τον γεωγραφικό αυτόν εντοπισμό καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά με τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Ορισμένοι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αναφέρονται στο αποτύπωμα άνθρακα. Θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να γίνει μια διάκριση και ενδεχομένως να πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε κάποια υλικά τα οποία προέρχονται από μια συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε για παράδειγμα κάποια υλικά τα οποία προέρχονται από πάρα πολύ μακρινές περιοχές χρησιμοποιούνται σε κάποια έργα, στο δικό μου το χωριό για παράδειγμα, περνάει ένας-δύο και στη συνέχεια πρέπει να αντικατασταθούν τα υλικά αυτά γιατί ουσιαστικά δεν ανταποκρίνονταν στις συνθήκες. Φαντάζομαι πάντως ότι σε σχέση με αυτό θα υποβληθούν τροπολογίες όσον αφορά την διάκριση α και β. Και η κυρία Ρούλε αναφέρθηκε σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει όντως εδώ πέρα μία διάκριση, η οποία γίνεται σε σχέση με την αρχική πρόταση. Είμαι πάντως αρκετά ευέλικτος. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να έχουμε πιο ευέλικτους κανόνες, ιδίως όσον αφορά την αγορά, παροχής νομικών υπηρεσιών ε, κτλ. ή όσον αφορά τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες στις οποίες αναφερθήκατε. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αμοιβαιότητα. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να αναφελεί να ανοίγει τις πόρτες της σε όλες τις αγορές, οι οποίες τελικά υποφελούνται της ελεύθερης αγοράς. Δεν αναφέρομαι στην Κίνα, αναφέρομαι και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ισχύει αυτή η αρχή της αμοιβαιότητας. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Ντεγκιούχτ, η Επίτροπη Ντεγκιούχτ και Μπαρνιέ ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να καταλήξουν σε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά την αμοιβαιότητα και όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών μας. Εμείς ανοίγουμε τις αγορές μας αλλά δεν κάνουν το ίδιο πράγμα και οι εταίροι μας πάντα. Πιστεύω ότι από νομικής πλευράς όντως θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε έννοιες. Κοιτάξτε, συνήθως λειτουργώ με τρόπο ιδιαίτερα πρακτικό. Ο κύριος Κρόιτσμαν αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Θα ακολουθήσω την σειρά τώρα των ομιλητών και δεν θα καταφέρω να απαντήσω δυστυχώς όλες τις ερωτήσεις. Πάντως μπορούμε και διμερώς να διευθετήσουμε κάποια ζητήματα και προφανώς θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσει στο μέλλον. Απλούστευση των κανόνων. Προφανώς όλοι το επιθυμούμε αυτό. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε όμως απλούστευση και απλοϊκότητα. Όταν λέω ότι θα πρέπει να πάμε προς τη χαμηλότερη τιμή, αυτό το οποίο λέω ουσιαστικά είναι ότι ε, έχουν οριμάσει πλέον τα πράγματα προκειμένου να καταφέρνουμε τελικά να χρησιμοποιούμε περισσότερο το μήτε, δηλαδή την πλέον συμφέρουσα οικονομικός προσφορά. Και βέβαια στην περίπτωση αυτή η τιμή θα είναι ένα σημαντικός παράγοντας και η τιμή στη τελευταία ανάλυση πάντα θα αποτελεί ένα σημείο αναφορά, ένα σημείο εκτίμηση. Μπορούμε σαφώ πάντα να δούμε την ποια καινοτόμα λύση, την τεχνικά καλύτερη λύση. Αν όμω είναι τρει-τέσσερι φορέ πιο ακριβή λύση αυτή, προφανώ δεν θα την εφαρμόσουμε. Η τιμή λοιπόν θα αποτελεί πάντα κριτήριο. Θα εξαρτηθεί όμως τώρα από το αν η υπηρεσία, το προϊόν είναι τυποποιημένο ή όχι, αν υπάρχει μια έντονη διάσταση καινοτομία κτλ. Με βάση τα κριτήρια αυτά θα βαρύνει περισσότερο ή λιγότερο και ο παράγοντας τιμή. Άκουσα τον κύριο Βάντεν Κάμπα που μίλησε και εξ ονόματος του κυρίου Έγκελ. Βλέπουμε ότι ε, η γενικότερη τάση είναι να καταφέρουμε να επηρεάσουμε περισσότερο την, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα έργα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν υπάρχουν τα απαραίτητα εργασιακά κοινωνικά κριτήρια όσον αφορά την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας κτλ. Μιλάμε για ανοιχτή αγορά, για μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμερίζουμε τις συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό το λόγο αναφέρομαι και σε μία διαδικασία που έχει να κάνει με την βιώσιμη παραγωγή και μας υποστηρίζει και το δικαστήριο στο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι στις 11 ή στις 10 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέληξε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση όσον αφορά τις κάτω χώρες και αναφέρθηκε στην, στο δίκαιο εμπόριο και στην ανάθεση μιας αγοράς. Τώρα για την υπεργολαβία. Ξέρω ότι τόσα προβλέπονται εδώ πέρα είναι αρκετά αυστηρά και άκαμπτα. Πάντως, ε, η υπεργολαβία μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέροντα μηχανισμό για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά παράλληλα συχνά αποτελεί και το είπε και αυτό και ο Σέρτζο Κοφεράτη, πηγή εγκληματικών ενεργειών, συμμετοχής δηλαδή εγκληματικών ενεργειών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε με τον πιο σαφή τρόπο την υπεργολαβία. Αν συνεργαζόμαστε, αν αναθέτουμε σε μια βασική Κύριε επιχείρηση που σε έναν δεύτερο, τρίτο, τέταρτο υπεργολάβο και εκεί πέρα φτάνουμε ουσιαστικά στη συμμετοχή μιας οργάνωσης παράνομης ή μιας εταιρεία που χρησιμοποιεί παράνομους μετανάστες για παράδειγμα, όπως για παράδειγμα είδαμε με μια ανάθεση βελγικής εταιρεία για τον καθαρισμό των σταθμών, είδαμε ότι στην περίπτωση αυτή υπήρχε η απασχόληση Παράνομο μεταναστών, οι οποίοι εργάζονταν σε πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το βλέπουμε και στη Γαλλία. Έγινε μια καταγγελία από την ΕΝΤΕΦ. Στην Φλομονβίλ, υπήρχαν Πολωνοί εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονταν χωρίς καμία προστασία στον τόπο εργασίας και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματο δεν υπάρχει καμία αποζημίωση και πρέπει απλώ να καταλήψουν τη δουλειά και να επιστρέψουν στα σπίτια του. Νομίζω λοιπόν ότι η υπεργολαφία θα πρέπει να εξυγιανθεί και θα πρέπει αυτό να γίνει με τρόπο αποτελεσματικό προκειμένου η εργασία, η ανάθεση τη δουλειά να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κοπεί τελικά την αναθέτουσα αρχή. Κύριε Κρότσμαν, το είπαμε και χθε. Επιμείνατε όντω στην στο ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ σαφείς ε, συγκεκριμένες προτάσεις. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ προσπάθησα να δω σχεδόν όλους αυτούς τους 75 ε, stakeholders, τα ενδιαφερόμενα μέρη που θέλαν τελικά να με συναντήσουν. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εθνική νομοθεσία, τις λογικές συμβάσεις και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε περισσότερη γραφειοκρατία. Χρειάζεται όμως μια ελάχιστη νομοθεσία και θα πρέπει να τηρεί την νομοθεσία αυτή και να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εφαρμόζεται. Για τα κριτήρια εξαίρεση τώρα επέκτηνε ενδεχομένω την έννοια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναφερόταν σε εμφανή διαφθορά. Εγώ αναφέρθηκα εδώ πέρα και σε κάποια κοινωνικά κριτήρια και είπα ότι δεν μπορούμε να εργαζόμαστε βάσει κάποιων υπονοιών υποψιών, αλλά βάσει συγκεκριμένων συνθήκων που προκύπτουν από τις νομοθεσίες. Για το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μίλησα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σήμερα να προωθήσουμε περισσότερο την έννοια της πλέον συμφέρουσας οικονομικός προσφοράς. Τώρα, Όσον αφορά την ε, κατηγοριοποίηση αυτή για την ανάθεση, ίσως προχώρησα λίγο περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό γιατί πιστεύω ότι ο βασικός στόχος είναι η συμμετοχή στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Είδαμε ότι οι δημόσιες αυτές συμβάσεις αντιστοιχούν στο 19-20% του ΑΕΠ και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτές τις δημόσιες συμβάσεις. Νομίζω πάντως ότι η προτινόμενη διαδικασία ήταν ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αναφέρθηκε και στην αμοιβαιότητα κυρία Ρούλε τώρα. Ναι, ο κατάλογος των ε, τεχνικών ε, διευκρινήσεων και προδιαγραφών. Το έκανα αυτό προκειμένου τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Τώρα διάκριση ανάμεσα σε α και σε β. Για ποιο, για ποιο λόγο τη διατηρούμε. Ακολουθώ εδώ πέρα την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δικό σας όμως το παράδειγμα αν για παράδειγμα κάποιες υπηρεσίες διάσωσης ε, ζημιώνονται, ναι, τότε συμφωνώ μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δημιουργήσω μεγαλύτερη γρεθοκρατία για κάποιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα διασυνοριακές, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν πιο ευέλικτες. Μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω αυτό. Η υπεργολαβία μόλις μίλησε για το ζήτημα αυτό καταλάβατε ότι εδώ πέρα αυτό που θέλω να πετύχουν είναι μία εξυγίανση σε σχέση με χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία. Τα πράγματα είναι σαφώς πιο ξεκάθαρα σήμερα από όταν στο παρελθόν, μόλον ότι υφίστανται ακόμα κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Το καταλάβατε αυτό με τα ξεκάθαρα παραδείγματα που σας έδωσα. Δεν θέλουμε να έχουμε αυτά τα υπερβολικά φαινόμενα διαδοχικής, υπερβολικής υπεργολαφίας, όταν αυτή μπορεί να αποφευχθεί. Άρθρο 84. Εθνικές ε, αρχές. Ξέρω ότι πολλές, πολλοί δεν βλέπουν πολύ θετικό μάτι τα όσα λέγονται στο σημείο αυτό. Πιστεύω ότι εκεί πέρα που δεν υπάρχουν εποπτικές αρχές θα πρέπει να δημιουργηθούν. Και πολλές φορές έχουμε πολλέ διαφορετικέ εθνικέ αρχέ. Κάρα δεν υπάρχει εναρμόνιση. Πρέπει να πετύχουμε ένα επίπεδο εναρμόνιση. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε στρεβλώσει, ε, διαφθορά. Όπου δεν υπάρχουν λοιπόν υποπτικές αρχές θα πρέπει να δημιουργηθούν. Κατά αυτόν τον τρόπο το άρθρο 84 με την τροποποίηση αυτή, αυτό προωθεί ουσιαστικά. Στη Γερμανία είναι τα κρατήδια αυτά τα οποία είναι υπεύθυνα για τις εποπτικές αρχές. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί μια ομοσπονδιακή εποπτική αρχή. Στη χώρα μου οι περιφέρειες ασχολούνται με το ζήτημα αυτό. Ξέρετε ότι αν ζητήσουμε τώρα από το Βέλγιο να δημιουργήσει μια ομοσπονδιακή κεντρική εθνική αρχή θα χρειαστούν δεκάδες χρόνια. Κοιτάξτε πόσες μέρες χρειάστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ε, κύριε Κοσνόνη, νομίζω ότι ήδη σας απάντησαν άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν πολλά αρνητικά παραδείγματα. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν Πολωνοί ή Τσέχοι άνθρωποι από τη χώρα σας να έρχονται και να εργάζονται σε απαράδεκτες συνθήκες σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να εργάζονται σε καλές συνθήκες δεν μπορούν να πληρώνονται 6-7 ευρώ την ώρα, ότι μπορεί η πληρωμή αυτή να είναι καλύτερη από ό,τι στην Τσεχία, την Πολωνία, τη Λιθουανία αλλά δεν μπορούμε εμεί αντικειμενικά να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Αναφερθήκατε στην ταγωνιστικότητα. δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για την χωρίς χωρί στήριση των κοινωνικών κανόνων. Γιατί διαφορετικά ουσιαστικά θα αντιμετωπίζουμε ορισμένου ανθρώπου σαν ήταν ζωικό κεφάλαιο τελικά. προσβεύεται κάποιες συντηρητικές θέσεις, εγώ κάποιες προ, πιο προδευτικές. Είναι λογικό να διαφέρουν οι απόψεις μας. Ο κύριος Δε τώρα. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε θα μπορούσα να ολοκληρώσω στο σημείο αυτό, κυρία Πετικάινεν, να e-procurement, ε, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Δεν τον έπτυξα αρκετά. Θέλω να είναι υποχρεωτικό το σύστημα αυτό, αρκεί να υπάρχει απαραίτητη κατάρτιση για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή κατάρτιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις τοπικές αρχές. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούν να γίνουν οικονομίες μέσω του ηλεκτρονικού αυτού συστήματος και για τις αναθέτουσες αρχέ και για τι ε, επιχειρήσει από ό,τι έχω δει στην Πορτογαλία, στην Γαλλία, στη Γερμανία Έχουν ξεκινήσει κάποια τέτοια προγράμματα, με συγχωρείτε, έχουμε κάποιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, οι οποίες όμως θα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο συντονισμένο. Θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατές, προκειμένου οι πληροφορίες να διαχέονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορούν τις πληροφορίες αυτές να τις χρησιμοποιήσουν και οι επιχειρήσεις και οι αναθέτουσες αρχές. Όταν όμως ε, Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μέσα και μπορεί άμεσα μια επιχείρηση να δει ότι υπάρχει η προκήρυξη ενό διαγωνισμού με τρόπο ηλεκτρονικό, που να περιμένει να διαβάσει την προκήρυξη αυτή σε, ποια, σε κάποια επίσημη εφημερίδα. Θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό. Θεωρώ επίσης ότι το σχετικό κόστος είναι χαμηλό, 1.180 ευρώ. Ε, μια επένδυση ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν είναι κάτι τόσο δαπανήρο. για τον κύκλο ζωής τώρα νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το εισάγουμε. Στις τεχνικές προδιαγραφές θα μπορούσε αυτό να εξαρτάται από διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, αλλά προς την ε, διαδικασία της ανάθεσης ουσιαστικά κινούμε εδώ πέρα στο δρόμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχουν κάποια κοινωνικά κριτήρια επιπλέον γιατί περιβαλλοντικά κριτήρια υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα οικολογικά σήματα τα οποία χρησιμοποιούνται. Κυρία Σμπέρκερ, κριτήρια επιλογής. Η τιμή προφανώς ε, αποτελεί τμήμα της πλέον συμφέρουσας οικονομικός προσφοράς. Είτε είναι τυποποιημένη υπηρεσία ή όχι, ε, θα επηρεάζει αυτό και τον παράγοντα τιμή, την βαρύτητα της τιμής. Κύριε Ζημάν, πολλές ε, ερωτήσεις. Λοιπόν, είμαστε υπέρ των δικασιών που περιγράψατε, όμως ε, θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτό ότι πρέπει προφανώς να εργαστούμε για να ε, ενισχύσουμε από νομική σκοπιά τις διάφορες έννοιες, να μην είμαστε αόριστοι και να αποφύγουμε να ανοίξουμε την πόρτα στις δικαστικές προσφυγές και φυσικά όλοι θα πρέπει να εργαστούμε αυτό μείωση των προθεσμιών. Το έκανα μόνο για τις ηλεκτρονικές προμήθειες δημοσίες συμβάσει, γιατί εγώ μπαίνω στη θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα περάσουν στις ηλεκτρονικές προμήθειες. Θα πρέπει να αντιδράσουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο χρονό να διαβιβάσουν την προσφορά ε, με το email, με το χειδρομείο, αλλά πρέπει να σκεφτεί και κάποιο την προσφορά. Αν πρόκειται για μια πιο πολύπλοκη προσφορά για έργα, για πολύπλοκες υπηρεσίε. για αρχιτεκτονικά έργα, πριν το χάρη. χρειάζεται χρόνος ε, για την προσφορά. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αν παραπέψουμε στι αρχικέ οδηγίε του 2017 17 και 18, είναι απλώ για να μην αγνοήσουμε και να τονίσουμε ότι στι μικρέ επιχειρήσει. Ε, δεν υπάρχει πληθώρα προσωπικού και χρειάζονται όλο το χρόνο προς διαθεσή τους ε, για να σκεφτούν μια προσφορά και να υποβάλουν την καλύτερη δυνατή προσφορά. Γι' αυτό ήθελα μεγαλύτερες προθεσμίες. Τώρα, ε, τώρα μέι, όταν λέμε Μέι, είναι αλήθεια ότι αιτιολογείται ε, πολλές φορές ε, εγώ δεν θέλω να γενικεύω, αλλά γενικά προτιμώ το σαλ, γιατί είμαστε πιο σίγουροι. Γιατί όταν λέμε ΜΕΙ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Για το α και β μπήλης επίσης, ε, κύριε Κονφεράτη, σας ευχαριστώ για αυτή την εκτίμηση για την ε, πλέον ε, συμφέρουσα οικονομικός προσφορά. Δεν μπορώ να περιμένω λιγότερο βέβαια από σένα. Σας ευχαριστώ επίσης ε, και σας συνάδελφε που κυρία Κορέτσα Είναι το τέλος του τουρνουά, δεν ξέρω μεταξύ ποιου και ποιου, αλλά στις 5. Ξέρετε, έχουμε και μια δραστηριότητα που θέλουμε να παρευρεθούμε και χαιρετίζω και τους πολλούς φίλους για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Τώρα, για την ευελιξία και για τους καλλιτέχνες και για τα ε, άλλα επαγγελματά διανοητικού χαρακτήρα. Τώρα, ε, ήταν ε, η καλύτερη παρέμβαση της ε, κυρίας που έφυγε, κυρία Κοράτσα. Κυρία Βάιλερ, μάλιστα. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα, που απάντησες στον κύριο Κοστίνσαφ πριν από μένα στο Σνούσιντ. και εγώ συμφωνώ με την πραγματικότητα που ανέφερε, κυρία Γκέμπαρτ, αξιότιμη δουλειά. Το σημείωσα αυτό. Αξιόλογη δουλειά, με συγχωρείτε. Αλλά όπω ήθελα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα ξεκινάει η δουλειά και έχουμε και την κατάθεση των τροπολογιών. Δεν ξέρω αν εξαρτάται από μένα, αλλά εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να έχουμε μεγαλύτερε προθεσμίε. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύπλοκο ο φάκελο αυτό, ότι θα έχουμε πάρα πολλέ τροπολογίε για τι προτάσει που έκανα και για ολόκληρε παραγράφου που δεν έχω αγγίξει καθόλου. Ακόμη και τι θα έχουμε τροπολογίε και είναι δύσκολο την εβδομάδα του Στρασβούργου να εργαζόμαστε σε επί διάφορων φακέλων, γιατί τρέχουμε από συνεδρίε σε συνεδρίε στο Στρασβούργο και σε ό,τι με αφορά αν αυτό αποφασιστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών, δηλαδή να έχουμε περαιτέρω προθεσμίε, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Σα ευχαριστώ για την καλή σα πρόθεση και για τη ε, διάθεσή σα να συνεχίσουμε τη δουλειά, γιατί από ό,τι φαντάζομαι θα συνεχιστεί ακόμη για μερικού μήνε. Ευχαριστώ, Μάρκα, για εξαιρετική δουλειά και για την εξαιρετική συζήτηση. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ, επειδή με πάθος και φλόγο υπεράσπισες το ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν είναι κατασυμβιβαστό με τον καλύτερο ανταγωνισμό το αντίθετο μάλιστα, αλλά ε, φαίνεται να υπάρχει και μια ιδεολογική απόκληση εδώ σε αυτό το φάκελο. Έτσι λοιπόν έχουμε λίγο χρόνο να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε κάπου αυτό το χάσμα. Αυτή την απόκληση, κατάθεση τροπολογιών 14 Ιουνίου, αυτή είναι η προθεσμία. Θα συζητήσουμε στις 9 και 10 Ιουλίου τις τροπολογίες, όμως νομίζω ότι θα συζητήσουμε και στους συντονιστές το θέμα της προθεσμίας. Σας ευχαριστώ και θα ξαναδώσω την Προεδρία στον κύριο Μάλκοπ Χάρμπορ. Uh, Κυρίε και κύριοι, περιμένει ο κύριο Κομφεράτη υπομονετικά. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Τραμπέλα για τη δέσμευσή του στο φάκελο αυτό. Αλλά έχει δίκιο, θα έχουμε μικροσκελή συζήτηση στο μέλλον και βεβαίω θα συζητήσουμε και το θέμα τη προθεσμία ε, για την κατάσταση τροπολογιών στη συνεδρία των συντονιστών σε λίγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι δεν μένετε για το τελευταίο σημείο, σας παρακαλώ αποχωρήστε με ησυχία από την αίθουσα για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Έτσι λοιπόν, θα εξετάσουμε τώρα το σχέδιο κειμένου του κυρίου Κοφεράτη σε σχέση με την ατζέντα για παρκής ασφαλής και βιώσιμες συντάξεις. Η κυρία Πετικάινεν γιατί κανεί είναι για το ΕΛΚ, ο κύριο Κρόιτσμαν ε, θα επανέλθει φαντάζομαι. Φεύγει ο κύριο Κρόιτσμαν. Μήπω θα επανέλθει γρήγορα. Η κυρία Τούρνεν είναι εδώ. Ο κύριο Τερτσίκ ε, δεν είναι εδώ, ο κύριος Δεγιόνκ είναι εδώ. Έχουμε λοιπόν ε, αρκετού από του σκιώδες. Κύριε Κονφεράτη, έχουμε καθυστερήσει λίγο με το χρονοδιάγραμμα, αλλά μπορείτε να μα παρουσιάσετε μια σύνοψη τη γνωμοδοτησής σα και κατόπιν θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου για να συνεισφέρουν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. έχουμε λίγους λοιπόν ηρικούς συναδέλφους ε, που ε, μπορούσαν να αντισταθούν στον καταιγισμό του κυρίου Ταραμπέλα. Ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους ε, για την εκθεσή μου σε πρώτερο στάδιο, αλλά επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, δεν θα αναφέρω τα πλήρη στοιχεία που γνωρίζουν οι συνάδελφοι και που έχουν σχολιάσει. Απλώ θέλω εντάχει να προσθέσω ορισμένες σκέψεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο κείμενο, το οποίο θα τροποποιηθεί στη συνέχεια. Τώρα, το πρώτο πρόβλημα που θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να προσθεθεί στο κείμενο αυτό είναι αυτό που αφορά μια ιδιαιτερότητα που μπορεί να εντοπιστεί στην εργασία πολλών ατόμων ε, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ε, η τάση, όπως είναι γνωστό, και που βασίζεται και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, να επιμηκύνεται ε, η εργασιακή ζωή των ατόμων και έτσι να απομακρύνεται η στιγμή της ταξιδότησής τους. Όμως τα άτομα που εργάζονται δεν εργάζονται όλα υπό τις ίδιες συνθήκες. Υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα, ε, κυρίως στο βιομηχανικό τομέα και στον ε, τομέα των, της μεταποίησης, που έχουν ένα χαρακτήρα πραγματικά φθοράς. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να εξετάζουμε με τον ίδιο τρόπο για να δώσω ένα κοινότυπο παράδειγμα. Πρέπει να το σε μια επιχείρηση συντηρουργίας ε, να θεωρούμε ε, ότι ένας τεχνικός που εργάζεται σε ένα γραφείο με air condition, ότι κάνει την ίδια δουλειά με έναν εργάτη που δουλεύει μπροστά ε, στην υψηκάμινο. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να υπάρχει και μία αντιστάθμιση η, το είδος της εργασίας με τα συστήματα συνταξιοδότησης. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη για να είμαστε δίκαιοι. Και γιατί πέρα από το παράδειγμα που έδωσα, Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το πόσο βαριά είναι η κάθε εργασία. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο σύστασης, γιατί και εδώ πρέπει να δώσουμε μια θετική απάντηση, στην αγορά εργασία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχει αυξηθεί η χρησιμοποίηση άτυπων συμβάσεων, δηλαδή έχουν προσθεθεί στην παραδοσιακή σύμβαση ορισμένου χρόνου, αρίστου χρόνου, κάποιες συμβάσεις ε, ορισμένου χρόνου, εποχικές συμβάσεις, εποχικές δραστηριότητες κτλ. Το σύστημα της ε, κεφαλαιοποίησης ε, μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, προστίθεται στο συμμετοχικό σύστημα. Ε, τα κενά που δεν καλύπτονται είτε από τη δραστηριότητα είτε από ε, την έλλειψη συνεισφορών είναι κάτι που δεν μπορούμε να ανακτήσουμε. Δηλαδή, για ένα άτομο που πολλάκις ε, υλοποιεί μια δραστηριότητα δυνάμει σύμβαση ορισμένου χρόνου στην εργασιακή του διαδρομή θα έχει κάποια κενά ε, σε ό,τι αφορά τις ε, ασφαλιστικές εισφορές και αυτό θα έχει αντίκτυπο στην τελική σύνταξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί σήμερα οι περισσότεροι νέοι αρχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέσω μιας ε, πρόσβασης στην εργασία που δύσκολα δίνεται από μια συμβασία ορίστου χρόνου σχεδόν πάντοτε βλέπουμε να υπάρχει επανάληψη άτυπων συμβάσεων. Τρίτο πρόβλημα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε ορισμένε ε, είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο, έχουμε κάποιες μορφές εργασίας παράνομης που υλοποιείται από άτομα που δεν έχουν ευρωπαϊκή υπηκότητα. Έτσι λοιπόν εργάζονται χωρίς να ισχύει για αυτούς ε, καμία σύμβαση και καμία νομοθεσία κάτι που κάποια στιγμή κάποτε λεγόταν μαύρη εργασία, σήμερα έχει αυτή την ε, περαιτέρω ε, συνιστόσα, γιατί ε, αυτή η παράνομη εργασία σήμερα στην Ευρώπη γίνεται από ανθρώπους που δεν είναι Ευρωπαίοι και δεν έχουν ευρωπαϊκή υπηκότητα. Έτσι λοιπόν ε, το επιβαρυντικό συστατικό είναι ότι τα άτομα αυτά, ε, για τα άτομα αυτά δεν δίνονται εισφορές. Και η αύξηση αυτού του είδους της δραστηριότητας ε, ουσιαστικά ε, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την ποιότητα της ζωής των ατόμων αυτών για το μέλλον, αλλά υπάρχει και κίνδυνος για το σύστημα. Έτσι λοιπόν υπάρχει ε, αποφυγή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως και αποφυγή για δύο λόγους. Η δραστηριότητα των ατόμων αυτών, ε, στο οποίο δεν αντιστοιχεί μια τελική σύνταξη, ε, ουσιαστικά ζημιώνει τελικά το συνταξιδετικό σύστημα, το σύστημα πρόνοιας. Και το άλλο σύνολο προβλημάτων έχει να κάνει με τη μεταβιβασιμότητα των συντάξεων. Σήμερα εμείς βλέπουμε μία σειρά ατόμων που εργάζονται, ε, καταβάλουν κάποιες εισφορές και κατόπιν επιστρέφουν στη χώρα τους. Όμως πλέον δεν έχουμε ε, τις ίδιες μεταναστευτικές διαδικασίες που είχαμε στο παρελθόν. Σε όλες τις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης ήταν ε, νορμάλ να έρχονται άτομα από τη Βόρεια Αφρική και στη συνέχεια να ζουν την υπόλοιπη ζωή τους ε, στην Ευρώπη. Όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα. Ε, στη Βόρεια Ευρώπη όπου οι χώρες των προσοβητικών κρατεών ε, δίνουν ε, πολύ εργατικό δυναμικό το ίδιο ισχύει και για την Νότια Ευρώπη έχουμε άτομα που προσφέρουν εργασία και έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην Αφρική και στην Ασία και στη συνέχεια όταν τα με αυτά επιστρέφουν στην πατρίδα τους ε, θα πρέπει να μπορούν να πάρουν ε, την ε, σύνταξη που κέρδισαν εργαζόμενοι εδώ. Έτσι λοιπόν χρειάζονται διασυνοριακοί κανόνες για να εγγυθούμε τους κανόνες αυτούς θα πρέπει να φανταστούμε όπως ε, τέθηκε και εγώ συμφωνώ με αυτή την πιθανή λύση, μία οδηγία, δηλαδή την κατάρτιση ε, μία οδηγία για ε, τις ε, οντότητες πρόνοιας, γιατί θα πρέπει να έχουν αυτές οι οντότητες, αυτή ακριβώς τη συγκεκριμένη εντολή και θα πρέπει να προβλέπουν και τη δυνατότητα μίας διαχείρισης της δραστηριότητάς τους πρόνοιας, που δεν αφορά μόνο τους κατοίκους, που διαμένουν, τους πολίτες που διαμένουν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία συνιστόσα διασυνοριακή, να καλύπτονται και μετανάστες δηλαδή. Αυτό το είχα εκφράσει την ε, περασμένη φορά και προκύπτει αυτό και από κάποιες σκέψεις που κάναμε γύρω από το ζήτημα φυσικά. Είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση θέλετε να μου υποβάλλετε μέσω τροπολογιών ε, για να ενισχύσουμε το συνολικό κείμενο. Uh, thank you very uh. Ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ σημαντικά αυτά σημεία για τις πλήρεις παρατηρήσεις που υποβάλατε. Ας ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις, κυρία Πέτικαν. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις πολύ καλές αυτές παρατηρήσεις και την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Δύο-τρία σημεία. Πρώτον, ναι, όντως θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις ε, μεθόδους ε, εκείνες που θα πείσουν τους ανθρώπους να μείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας, γιατί αυτό αποτελεί σημαντικό ακρογωνιαίο λίθο της ε, σταθερότητας του συνταξιωτικού μας συστήματος και των συνταξιωτικών ταμείων. Κοινή βέβαια είναι η ευθύνη εδώ πέρα και των ίδιων των εργαζομένων και των εργοδοτών και του δημοσίου τομέα. Ο εισηγητή επίσης αναφέρθηκε σε κάποια επιμέρους σημεία τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Οι σύντομε περίοδοι εργασία στι οποίες αναφέρθηκες, πώς μπορούμε δηλαδή να διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε και συντάξεις για τις περιόδους αυτές. Τώρα, όσον αφορά την ηλικία ταξιοδότησης και με αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη μεταφορά των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων προκειμένου να μην αφαιρηθούν τα δικαιώματα αυτά από την σύνταξη που δικαιούται στο τέλος το άτομο αυτό. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση ενός ελάχιστου επίπεδου των συντάξεων και θα πρέπει να υπάρχει και μια σχετική εναρμόνιση των κανονισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρχει ένα λογικό επίπεδο στις συντάξεις. Υπάρχουν ε, πολλοί άνθρωποι που εργάζονται σε διάφορα κράτη-μέλη και για τους ανθρώπους αυτούς θα θέλαμε να θαρρύνουμε ένα ισότιμο σύστημα. Σίγουρα αυτό δεν είναι εύκολο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ταχθεί ε, υπέρ διαφόρων μοντέλων εναρμόνισης των συντάξεων. Ενδεχομένως να λοχεύουν κάποιοι κίνδυνοι βέβαια στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρουμε σε ποιο επίπεδο σύνταξη τελικά θα καταλήξουμε και αν θα υπάρχουν διαφορές από τον έναν εργαζόμενο στον άλλον με βάση το ποιο είναι εργοδότης ή ποια είναι η χώρα της απασχόλησης. Κάποιες ακόμα παρατηρήσεις. Συντάξεις για τις γυναίκες. Σαφώ οι συντάξει αυτέ θα πρέπει να τα αποκρίνονται στα χρόνια απασχόληση. Πολύ συχνά όμω ξέρουμε ότι οι γυναίκε έχουν χαμηλότερου μισθού και αναγκάζονται να μείνουν πιο συχνά στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά. Επομένω, καταλήγουν να έχουν και χαμηλού μισθού και χαμηλέ συντάξει στη συνέχεια. Πιστεύω ότι αυτό πολύ σοβαρά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν εξετάζουμε τα μοντέλα υπολογισμού των συντάξεων για τις γυναίκες. Και τέλος, Αλέξη, ίσως σημαντικό, ένα ζήτημα πολιτικές φύσης, πολιτικής φύσης. Όταν μιλάμε για την κρίση στον συνταξιδοτικό τομέα, πιστεύω ότι θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι οι συνταξιούχοι δεν αποτελούν βάρος στις κοινωνίες, αλλά είναι και πολύ σημαντικοί καταναλωτές. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σύστημα των συντάξεων της Ευρώπης πιέζεται όλο και περισσότερο και αυτό θα ενισχυθεί και στα επόμενα χρόνια. Οπότε χαιρετίζω την τοποθέτηση και γνωμοδότηση του κυρίου ο Κοφεράτη που καλεί την ε, Επιτροπή να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της αλλά δεν πρέπει να ξεχνήσουμε να αναφέρουμε τα προβλήματα και την οικονομική κρίση η οποία ενισχύει τα προβλήματα των συντάξεων και τις δημογραφικές αλλαγές διότι βλέπουμε ότι ίσως απλώς το οικονομικό σύστημα επηρέασε αρνητικά τη συντάξεις και θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες αποδόσεις και να υπάρχει μία δυνατότητα συμπληρώσεως των ε, ε, συντάξεων. Υπάρχουν εξαιρετικές, ε, εξαιρετικά ταμεία συντάξεως και πληρώνεται πολύ λίγο και σχετικά δίδουν υψηλές συντάξεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το εξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει διάφορα μέτρα, αλλά ουσιαστικά το θέμα είναι η, η ηλικία συνταξιοδοτήσεως και η ε, ο συσχετισμός τους με το προσδόκιμο ζωής διότι όσον αφορά την, την υποχρεωτική ή εθελοντική συνταξιοδότηση υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις και δεν μπορούμε απλώς να βασιστούμε εις τις προσδοκίες των ανθρώπων δεν μπορούμε να ε, έχουμε συνεχώς εξαιρέσει. Βέβαια στη Γερμανία συνέχεια ζητούνται εξαιρέσει και ε, τα βαρέα και ανθίγυνα ε, δεν μπορούν να εξασκούνται μέχρι τα 65 έτη αλλά από εκεί θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εμπλακούν. Αν δω πόσο πάλι ε, βρίσκουν ευέλικτα συστήματα στις συλλογικές συμβάσεις ε, με τις οποίες μπορεί κανείς να συνταξιοδοτηθεί πιο νωρίς πιστεύω ότι η λύση αυτή είναι η σωστή και αυτή θα έπρεπε να ακολουθήσουμε και εμείς και γι' αυτό και το επαναλαμβάνω υπάρχουν ε, συστήματα τα οποία είναι προφητικά για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μεταξύ των οποίων μπορούμε να προχωρήσουμε. Βέβαια δεν μπορούμε να γενικεύουμε όλες τις ε, αρχές αλλά χρειάζονται συλλογικές συμβάσεις. Ε, κύριε Κομφεράτη, ε, δεν έχω αντιληφθεί με τι χρήματα θα καταρτήσετε το σύστημά σας και πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο έχουμε προκλήσεις και είναι σαφές ότι ο σημερινός επαγγελματικός κόσμος διαφέρει πάρα πολύ από το παρελθόν. Εάν ε, θέλω να εργάζομαι 30-40 χρόνια βλέπουμε ότι οι δομές είναι διαφορετικές και δεν θέλουμε να φτάσουμε στα γεράματά μας στη φτώχεια και ε, πρέπει γι' αυτό να κάνουμε επιπλέον προσπάθειες και γι' αυτό θα χρειαστούμε χρειαστούν και ρυθμιστικές διατάξεις και εδώ αναφέρομαι το θέμα της ρευστότητος και της φερεγγιότητος των συνταξιοδοτικών συστημάτων διότι βλέπουμε αν υπάρχουν συστήματα αμοιβαίων ασφαλίσεων δεν έχω πρόβλημα αλλά δεν πρέπει πρέπει να προεξοφλεί ότι θα είναι φερέγγιες οι εταιρείε αυτές όταν συνταξιοδοτείται κάπως και ευχαριστώ τον εισηγητή. Κυρία Τούρανεν, ευχαριστούμε. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την, τον εισηγητή. Η μεγάλη αυτή συζήτηση για τις συντάξεις καλύπτει ουσιαστικά δύο βασικούς τομείς. το αν τελικά η σύνταξη αρκεί, προκειμένου να ζει κανείς με αξιοπρέπεια, και το δεύτερο ζήτημα είναι η βιωσιμότητα του συνταξιδοτικού συστήματος. Στη μεγάλη αυτή ευρεία συζήτηση εμείς ε, οι πράσινοι έχουμε μία κοινή θέση. Λέμε ουσιαστικά ότι ε, είμαστε υπέρ μεταρρυθμίσεων στο σύστημα το συνταξιδοτικό προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το συνταξιδοτικό σύστημα θα μπορέσει να αποκριθεί στις δημογραφικές αλλαγές, στην αύξηση προσδοκίμου ζωής, στην διαφοροποίηση της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει όμως οι συντάξεις αυτές να είναι δίκαιες και θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο στην αλληλεγγύη και όχι να βάλουν κατά της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η βασική μας κοινή προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως να θέσει ηλικία συνταξιοδότησης. Δεν νομίζω καν ότι έχουμε αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο. Επί της αρχής όμως, νομίζω ότι δεν θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αύξηση της ηλικίας εξοδότησης. Αυτό έχει γίνει ήδη αρκετά σε ορισμένα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει τώρα κατά προτεραιότητα. Ένα άλλο βασικό ζήτημα για μας είναι ότι είναι ο πρώτος πυλώνας. Είμαστε υπέρ ενός συστήματος με πολλούς πυλώνες, αλλά θα θέλουμε στον πρώτο πυλώνα να μπορούμε να προστατεύουμε ουσιαστικά του ανθρώπους από την ένδυα, από τη φτώχεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν επικουρικές επιπλέον συντάξεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η βασική σύνταξη που παίρνουν ως μόνη σύνταξη ορισμένοι άνθρωποι θα πρέπει να τους προστατεύει από τη φτώχεια κάποια ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν ιδιαίτερα τη δική μας τώρα την Επιτροπή. Να αυξήσουμε την διάσταση ίνκο της έκθεσης αυτής, δηλαδή τα δικαιώματα των συνταξιούχων ως καταναλωτών, καλύτερη πληροφόρηση και προστασία των δικαιωμάτων τους. Νομίζω και αυτό και άλλα κοινωνικά ζητήματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Στον δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα θα πρέπει να μπορέσουμε να υποβάλουμε κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις προς την, επιβολή απασχόλησης, προς την Επιτροπή Απασχόλησης, ιδίως κατά τη διάρκεια τώρα της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Θεωρούμε ότι ε, ο τρίτος πυλώνας έχει ζημιωθεί ιδιαίτερα. Ορισμένα συντοξιδοτικά ταμεία προχώρησαν σε πολλές επικίνδυνες ε, επενδύσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις έχασαν ακόμα και 30% ορισμένοι συνταξιούχοι 30% των αποταμιεύσεων τους, των συνταξιδοτικών τους αποταμιεύσεων. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε αυτού του είδους ε, την έκθεση σε κίνδυνο στο μέλλον. Και ένα ακόμα ζήτημα είναι ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε από τη σχετική ψηφοφορία την προηγούμενη εβδομάδα να αφήσει εκτός το ζήτημα των συντάξεων. Είναι πολύ σημαντικό να ισχύει ο φόρος αυτός και για τα συνταξιδοτικά ταμεία, γιατί δεν θα πρέπει να κάνουν μόνο βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να έχουν μια πιο μεγαλεπίβολη ενόραση του μέλλοντος. Δεύτερον τώρα, Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου οι επενδύσεις από τα εξωτικά ταμεία να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνε. Και ως προς αυτός πρέπει να κάνουμε ακόμα πολύ ακόμη δουλειά. Έχω εξετάσει το χρηματοδοτικό πορτοφόλιο, επενδυτικό πορτοφόλιο από διάφορες ε, διάφορα στα εξωτικά ταμεία, ιδιωτικού ιδιωτικούς εξωτικούς οργανισμούς από τη χώρα μου και πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και πληροφόρηση για τους καταναλωτές, ιδίως τον τρίτο πυλώνα, προκειμένου να μπορούν να λάβουν σωστά, σωστές αποφάσεις, να βασίζονται σωστές πληροφορίες. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα μεταφοράς των σταξιδικών δικαιωμάτων, ιδίως στον δεύτερο πυλώνα. Θα μπορούσαμε να απτύξουμε περισσότερο το σημείο 7. Δηλαδή, να δίνει τη δυνατότητα στους ορισμένους εργαζόμενους να, έχουν, να μεταφέρουν τα σταξιδικά τους δικαιώματα όταν πηγαίνουν σε έναν άλλον εργοδότη ή στο ενδιάμεσο διάστημα να μπορούν να έχουν ένα σύστημα, αν θέλετε, καταγραφή το οποίο να ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή πηγαίνοντας από τον εργοδότη στον άλλον να καταγράφονται σε ένα μητρό τα συνταξιωτικά τους δικαιώματα κεφαλαϊκές, κεφαλαϊκές απαιτήσει. Θα πρέπει και τα ιδιωτικά συντοξιδοτικά ταμεία να έχουν τα απαραίτητα διαθέσιμα κεφάλαια προκειμένου να μπορέσουν να αποκριθούν σε περίοδους οικονομικής κρίσης. Πιστεύω ότι ως Επιτροπή ΙΜΚΟ, τουλάχιστον από τη δική μου πολιτική ομάδα, πρέπει να θέσουμε αυτές τις τροπολογίες. Είμαστε υπέρ όμως των περισσότερων πραγμάτων που έχει ήδη πει ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ορθές παρατηρήσεις. Έχετε δίκιο. Σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτά τα σημεία και εγώ έχω κάποια σχόλια. Ο κύριος Δεγιόν καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σιγητή. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Αυτά που λέτε στο σημείο 3, κύριε Σιγητά, είναι πολύ θετικά. Κατά την άποψή μου, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μειώσουμε την ανεργία και για την κατηγορία ε, των εργαζομένων που βρίσκονται γύρω στα 55 έτη Στι κάτω χώρε, πρέπει χάρη οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Στην Επιτροπή ΙΜΚΟ δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των συνταξιωτικών ε, ταμείων. Ε, δεν είμαστε καθελήν αρμόδιοι, όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες συστάσεις. Επίσης, ε, στο δεύτερο πυλώνα, να πω ότι συμφωνώ με όσο υπόθηκαν από την κυρία Τουρούνεν, θα πρέπει ο πρώτος πυλώνας να είναι ο κύριος πυλώνα, αλλά ο δεύτερος πυλώνας ω συλλογική σύνταξη θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτό το ζήτημα. Και κατόπιν, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ ήδη μιλήσαμε για την αναγκαιότητα να αποσαφηνίσουμε την οδηγία που αφορά τις ε, κεφαλαϊκές απαιτήσει για τα εξοδοξιδοτικά συστήματα. Υπάρχουν ε, δύο κεφαλαϊκές απαιτήσει ε, που εφαρμόζονται, που ισχύουν για τα εξοδοξιδοτικά ταμεία θα πρέπει να πούμε κάτι για το θέμα αυτό αναλόγω και με το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Επίσης, την τελευταία φορά μιλήσαμε για την ε, δυνατότητα μεταφορά των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης. Ε, έχουμε δύο προβλήματα. Έχουμε και τις φορολογικές πτυχές Σίγουρα τα δικαιώματα, ε, το ότι οριμάζουν σε μια χώρα και θα πρέπει κάποιος να απολάβει αυτά τα δικαιώματα σε μια άλλη χώρα δημιουργεί κάποιες δυσκολίες, αλλά θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό. Και καθώς ε, υπάρχουν ε, διάφορες μορφές πρόνοιας, δυνάμει του δεύτερου πυλώνα, είναι δύσκολο ένα σύστημα συντοξιδοτικό που ε, είναι κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα να μπορεί να συνδυαστεί με ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα. Είναι λοιπόν δύσκολο να υπολογίσουμε τα συνταξιδοτικά δικαιώματα των ε, διάφορων συστημάτων πρόνοιας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δημιουργεί μία επιπλέον δυσκολία για τα συνταξιδοτικά ταμεία και πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να καταθέσει μία πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με τον υπολογισμό των διαφόρων ειδών συντάξεων. Εμεί πρέπει να το ζητήσουμε αυτό σε Επιτροπή ΙΜΚΟ. Και κατόπιν, μιλήσατε για ένα σύστημα καταγραφής, tracking, για να γνωρίζουμε τι είδου ε, σύστημα εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Και επίση ε, συμφωνώ με όσα είπε η κυρία Τουρνέρ για τον τρίτο πυλώνα. Δηλαδή, η χορήγηση πληροφοριών στον καταναλωτή για να γνωρίζει και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και επίση, ε, χρειάζεται να είμαστε σαφεί για το σε τι συνίσταται στην πραγματικότητα ο τρίτο πυλώνα. Για να ξέρουμε αν, παραδείγματο χάρη, κάποιο έχει πιο χαμηλή σύνταξη. Όλα αυτά δημιουργούν ε, σύγχυση και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Uh, and Mrs. final speaker. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση την οποία μόλις ακούσαμε απέδειξε ότι το σύστημα των συντάξεων στα κράτη-μέλη διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό και οι απαντήσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν είναι τελείως διαφορετικές. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε. Αυτό όμως το οποίο είναι σαφές είναι ότι για μένα η πρόταση του Σέτζιο Κοφεράτη ε, τονίζει ότι πρέπει να φροντίσουμε ο πρώτος πιλότητας να είναι ο πιο σημαντικός γιατί αυτός είναι που θα φροντίσει να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων ε, στην, ε, στα γερατιά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει μία σύνταξη από την επιχείρηση, δεν υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας και ο τρίτος πυλώνας είναι μία ιδιωτική ασφάλιση, αλλά ποιος μπορεί ε, να την σηκώσει. Κάποιος ο οποίος ε, ε, ε, είναι εύπορος αλλά όχι οι υπόλοιποι. Αυτοί που κάνουν μικροδουλίτσες στη Γερμανία οι οποίοι θεωρούν ότι ο καλός ακαθάριστος μισθός τους είναι 1000 ευρώ το μήνα. Αυτοί δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτα και αυτοί χρειάζονται ως επτοπλίστων αυτή τη σύνταξη και δεν μπορούν να την έχουν. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ο πρώτος πυλώνας είναι ο πιο βασικός. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που είπε ο σχετικά με την ηλικία συνταξιοδοτήσεως είναι πολύ βασικό. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι διότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειές που είναι σωματικά πολύ δύσκολες και βαριές και δεν μπορούν να δουλέψουν ε, μέχρι τα 65, μέχρι ε, τα 60 και πολύ. Και ορισμένοι οι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν ε, ψυχικό σθένος ε, αλλά και άλλοι πάλι οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν μέχρι τα 65 ή και τα 70 άρα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και όταν βλέπουμε ότι η ηλικία συνταξιοδοτήσεως ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι κάτω από τα 60 είναι μια τελείως ακαδημαϊκή συζήτηση εάν θα συζητάμε για 62 65 ή 67 διότι οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους στα 60 δεν πρόκειται να βρουν άλλη δουλειά και πρέπει να σκεφτούμε εάν δεν μπορούμε και στο δεύτερο πυλώνα να βρούμε ορισμένα κίνητρα και να δούμε εάν ο κύριος Κοφεράτη θα δεχθεί την ιδέα μου κατά τρόπον ώστε οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν ιδίως άτομα τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους πάνω από 55 ετών πρέπει να πληρώνουν και έκτακτη συνδρομή στα ταμεία για να μπορέσουν να δώσουν ένα επιπλέον εισόδημα στα άτομα αυτά. Πρέπει λοιπόν ε, να εμπλακούν περισσότερο και οι επιχειρήσεις. Είναι μια ιδέα που μου ήρθε εχθές και θα ήθελα να τη συζητήσουμε. Πιστεύω όμως και αυτό ελέγχθη ήδη, η κατάσταση των γυναικών είναι τέτοια ώστε πρέπει να την έχουμε υπόψη μας για διότι η φτώχεια στα γεράματα είναι ιδίως γυναικεία φτώχεια στα γεράματα και αυτό θα δούμε ότι δεν πρόκειται να επιληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χρειαστούν πιο σοβαρές επεμβάσεις κατά τρόπον ώστε να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ του εισοδήματος των ανδρών και των γυναικών και να μπορέσουν να προσεγγίσουν διότι έτσι μόνο θα λύσουμε και το πρόβλημα της φτώχειας στα γεράματα. Ευχαριστώ. Ε, επειδή δεν είναι ο σκιώδης εισηγητής μας μπορώ κάτι να προσθέσω διότι νομίζω ότι σε μία ώρα θα τελειώσουμε τις δουλειές μας. Καταρχήν, σχετικά με ορισμένους τομείς ε, που ανησυχούν ε, τους πολίτες στην ενιαία αγορά. Ε, είναι, είναι από τα μεγαλύτερα μελήματα των εργαζομένων το θέμα της σύνταξής τους και ε, το θέμα του πυλώνα μας απασχολεί. Σχετικά με το πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 είναι ότι το να βασίζεται κανείς ορισμένες χώρος ε, σε μία σύνταξη του πυλώνα ε, τους ε, έχει δέσμιους και δεν μπορούν να μετακινηθούν και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε να κινηθούν για να αναπτύξουν τις καριέρες τους θα θέλαμε και εμείς να μπορέσουν να καλύψουν και άλλες δυνατότητες ε, και αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό γι' αυτό και η Γενική Διεύθυνση ε, της Ερευνάς ε, σκέφτεται να καταρτήσει ένα χωριστό σύστημα συνταξιοδοτήσεως των ερευνητών και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα μειονέκτημα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει και την μισή τους καριέρα στο δημόσιο και τη μισή στον ιδιωτικό τομέα. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, για την ευρωπαϊκή οικονομία και θα πρέπει να δούμε ε, ως θεματοφύλακες της ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες ότι υπάρχουν πραγματικά ορισμένα προβλήματα τα οποία μειώνουν τις δυνατότητες ορισμένων πολιτών ε, και αναφέρομαι εδώ στο σύστημα των Ιταλικών συντάξεων που είναι ίσως ενδιαφέρον διότι ένας πολίτης της περιοχής μου ο οποίος εργάστηκε μία δεκαετία στην Ιταλία έπαθε μία πάθηση στο μάτι, χρειάστηκε ε, να πάρει σύνταξη αναπηρίας την οποία ε, ζήτησε όταν εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μπορούσε να την πληρωθεί και το σύστημα Solvit στην Αγγλία του, τον δικαίωση. Προσπάθησε επί ένα χρόνο να πείσει τους Ιταλούς να τον πληρώσουν και έξι μήνες αφού εστράφει στο Σόλβιτ άρχισε να παίρνει τη σύνταξή του. Οπότε βλέπετε ότι είναι άτομα που έχουν δικαιώματα στον πρώτο πυλώνα και θα έπρεπε εδώ στην Επιτροπή μας να δούμε ότι είναι πολύ καλή ιδέα αυτή να υπάρχει μια ανταλλαγή πληροφοριών αλλά είναι σαφώς ότι το Solvit υπάρχει για να λύσει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας και καλό θα ήταν ε, κάτι να λεχθεί στα πλαίσια αυτά. Σας ευχαριστώ. Ε, δεν νομίζω ότι είναι κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και τώρα ο κύριος Κοφεράτη μπορεί να κλείσει σύντομα για να ξεκινήσουμε 5.30 την συνεδρίασή μας. Έχετε δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για όλες τις σκέψεις ε, και τις προτάσεις που προσέθησαν εδώ σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Θέλω να πω όμως ε, και λίγα πράγματα. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νομοθετική αρμοδιότητα για τα συνταξιδοτικά. Αρμοδιότητα έχουν ε, τα κράτη-μέλη. Εμείς απλώς πρέπει να αναφέρουμε κάποια κριτήρια που θα μας οδηγούν σε μια επιθυμητή ομοιογένεια του συστήματος και να προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε τη σταθερότητα των συνταξιδοτικών συστημάτων, όπως λέει και ο τίτλος, και ε, για το λόγο αυτό εμείς μαζί με τις υπόλοιπες επιτροπές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα σε σχέση με το τι έγινε ακόμη και στα πλαίσια της, της πρότασης της Λευκής Βίβλου. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν ε, μίλησα εκτενώς για το θέμα αυτό γιατί το είχα την περασμένη φορά. Είμαστε ενώπιοι ενό προβλήματο που μπορεί να γίνει δραματικό για εκατομμύρια ανθρώπου στην Ευρώπη. Όλε οι χώρε ε, περνούν ε, από συνταξιδοτικά συστήματα που ήταν ε, συμμετοχικά συστήματα σε συστήματα κεφαλαιοποιητικά. Οι γυναίκες έχουν τη μητρότητα, έχουν αναλάβει τη θεραπεία της φροντίδα και αμείβονται, όσο, και αμείβονται λιγότερο. Και βλέπουμε ότι ο κυκλό ε, κλείνει δραματικά γιατί υπάρχει ο κίνδυνο να συνταξιδοτηθούν δυνάμει συνθήκων που κατόπιν ε, θα τι επιβαρύνουν για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που ε, μπορούμε εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει εκ των προτέρων να παρεύουμε για τα συνταξιδοτικά συστήματα και τα συστήματα Γι' αυτό επιμένω για το βάρο του πρώτου πυλώνα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αξία του δεύτερου και τη χρησιμότητα του τρίτου πυλώνα, όμω εμεί δεν ε, θα κατορθώσουμε να δώσουμε μια θετική προοπτική σε κανέναν αν δεν είναι κατάλληλος ο πρώτος πυλώνας και αν δεν εγγυείται, δεν εγγυάται σε εκατομμύρια άτομα σε 30-40 χρόνια να ε, μπουν σε κατάσταση φτώχεια. να αποφύγουν να μπουν σε κατάσταση φτώχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρογνωμοσύνη σα και για το θέμα αυτό. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 12 Ιουνίου στι 12 το μεσημέρι. Θα εξετάσουμε τι ε, τροπολογίε, θα ψηφίσουμε